Ξεκινάμε λοιπόν τη συνάντηση της Επιτροπής μας και σας παρακαλώ στις θέσεις σας. Επαναλαμβάνω στις θέσεις σας. Ακούγεται το μικρόφωνο μου, ρωτάει ο Πρόεδρος. Και βέβαια ακούγεται. Παρακαλώ λοιπόν στις θέσεις σας. Prego di prendere posto. Παρακαλώ για πολλωστή φορά να επαναλάβω στις θέσεις σας. Sono stato col tuo ministro stamattina. La barra. Allora, approvazione dell'ordine να εγκρίνουμε, τα πρακτι... να την ημερήσια διάταξη. Δεν ακούμε κάποια παρατήρηση, αλλά λοιπόν εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έγκριση τώρα των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας 20-27 Οκτωβρίου. Εγκρίνονται και εδώ τα πρακτικά. Να ευχηθώ σε όλους το καλώς ήλθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη σημαντική αυτή μερίδα εργασίας για την κατάσταση των νέων γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε αυτό το σεμινάριο για την κατάσταση των νέων αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι αποτελεί από τα θέματα τα περισσότερο σημαντικά στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουμε ένα κίνδυνο ότι το φαινόμενο της γύρασης αντιμετωπίζουμε και κίνδυνος για τη γεωργία. Πολλοί γεωργοί θυμούνται ότι μόνο το, 20, μόνο το 7% είναι νεότεροι των 35 ετών Ευρωπαίοι γεωργοί και 24,5 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι γεωργοί θα συντοξιδοτηθούν τα επόμενα 10 χρόνια και από την έκθεση Περάλντι για το μέλλον των νέων γεωργών και συνεχίζοντας με τον George Lyon για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013 έχουμε την Επιτροπή μας που τόνισε ότι απαιτούνται μέτρα και αυτό για να υποστηρίξουμε τους νέους στη γεωργία μέσω των πριν εγκατάσταση επιδοτήσεων εγκατάσταση και επιδοτήσει υποδικίου για την εγκατάσταση, όπως επίση κάποιες παροτρήσει μέσω ε, των ε, ταμείων ε, των κονδυλίων του δευτέρου πυλώνα. Η πρόσφατη ανακοίνωση τη Επιτροπή για την Γενική Γεωργική Πολιτική το 2020 ότι θα πρέπει να αποκριθούμε στι απαιτήσει για τους νέους γεωργούς και ελπίζουμε όλα αυτά να μεταφραστούν στην πραγματικότητα όσο γίνεται πιο σύντομα. Για, τη σημερινή... για το σημερινό απόγευμα εργασία. Ε, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα προσκαλέσαμε δύο εμπειρογνώμενες, την κυρία Αλντόμαν Τζαβόισκα από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας που θα ήθελα να χαιρετήσω και να ορίσω ένθερμα από πλευράς Επιτροπής μας το Σταξμπιστ από το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ δυστυχώς λόγω ε, προβλημάτων καιρού παρέμεινε στην Αγγλία δεν μπόρεσε να έλθει και δυστυχώς λυπάμαι και για άλλους συναδέλφους που δεν τα κατάφεραν να έλθουν μέχρι εδώ ακριβώς επειδή βλέπουμε τις ε, μετρολογικές συνθήκες. Επίσης ε, το πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Προεδρείου. Θα ήθελα εδώ από το ΣΕΖΑ και δω το λόγο στην εμπειρογνώμονά μας και στη συνέχεια βέβαια θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από το Γιώρης Μπάκλα τη ΣΕΖΑ, τον πρόεδρο. Η κυρία Αλντόνα Σαβοσκα έχει το λόγο. Δυσκολευόμαστε στο να ανοίξουμε το μικρόφωνο της κυρίας. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε θέση και μικρόφωνο. Υπομονή, υπομονή να λύσουμε το πρόβλημα το τεχνικό του μικροφόνου. Εντάξει, λειτουργεί τώρα. Όλα καλά. Ε, mm, Αγαπητέ Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των νέων γεωργών και όλων των νέων που ζουν στις αγροτικές περιοχές, Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έκθεσής μου η οποία μου ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών που αφορά την κατάσταση των νέων παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο στόχος ήταν να προτείνουμε μερικές ε, να παρουσιάσουμε μερικέ προτάσεις για βελτίωση των αδυναμιών και λήψεων. Ε, και πράγματι είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω αυτό το έργο διότι έχω παρακολουθεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ε, συζητήσεις, έχω ενημερωθεί για τις πρόσφατες έρευνες, ε, για τα στοιχεία της γεωργίας, του αγροτικού τομέα και είμαι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα προβλήματα ε, που διαπιστώθηκαν στις ε, νέες χώρες, δηλαδή στις ε, χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ε, ξέρουμε όλοι, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πολλές προκλήσεις, αλλά παρουσιάζει και θαυμάσιες ευκαιρίες, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα από την Πολωνική Γεωργία. Πριν από την ένταξή μας δεν καλύπτονταν από τόσο μεγάλη κρατική βοήθεια όσο καλύπτονται τώρα μετά την ένταξη. Επίσης, ε, ε, ε, εγώ δεν είμαι νέα παραγωγός και δεν καλύπτουμε από τις διατάξεις, αλλά κατανοώ πλήρως την θέση των νέων αυτών παραγωγών και ιδίως όσους θέλουν να αρχίσουν μια να ασχολούνται σε αυτόν τον παραγωγικό τομέα. Θέλουν να ξεκινήσουν μια αγροτική εκμετάλλευση ή μια μονάδα αγροτική. Λοιπόν, η έκθεσή μου παρουσιάζει πολλά στατιστικά στοιχεία, πίνακες, γραφήματα. Καταρχάς, γενικά, πρέπει να πω ότι η παρουσία νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα Α, ε, όχι, επαναλαμβάνω τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί είναι δικαιολογημένα στον αγροτικό τομέα, διότι η Ήπεθρος παρουσιάζει μια γύρανση του πληθυσμού και πολλοί νέοι δεν βρίσκουν απασχόληση και αναγκάζονται να φύγουν από την Ήπεθρο και να πάνε στα αστικά κέντρα για να βρουν δουλειά. Εγώ ασχολήθηκα κυρίως με τα δεδομένα, με τα στοιχεία νέων παραγωγών, αλλά Ορισμένα συμπεράσματα συμπίπτουν και με τις τάσεις του γενικού πληθυσμού. Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι όταν αναφερόμαστε σε χρήστες ή ιδιοκτήτες αγροτικών μονάδων η τάση που διαγράφεται είναι πτωτική Δηλαδή μειώνεται ο ρυθμός των νέων απασχολούμενων διότι όπως είπαμε μετακινούνται σε αστικά κέντρα παρόλο που μπορεί να προέρχονται από αγροτικές οικογένειες. Όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε περίπου 233 νέους παραγωγούς που ήταν ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων και 4,5 εκατομμύρια ε, παραγωγών ε, ηλικίας 65 και άνω. Δηλαδή είχαμε μόνο 6% νέων κάτω των 35 και 34% των παραγωγών που ήταν πάνω από 65 ετών. Βεβαίω αυτά στα στοιχεία θα ήταν καλύτερα εάν είχαμε συνυπολογίσει και την ε, χρήση αγροτικής γης από νέους ανθρώπους. 8% των νέων ε, το, καλλιεργούσαν 8% ε, της αγροτικής έκτασης, 8,6% του καλλιεργούσαν νέοι παραγωγοί και 14% μεγαλύτερης ηλικίας. Εδώ βλέπετε τους ιδιοκτήτες αναηλικία. Και βλέπετε μια σημαντική μείωση του αριθμού των ιδιοκτητών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ νέων αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αυτή η μείωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν 36%. Ήταν μικρότερη η μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15% όπου ο ορισμός των νέων ε, παραγωγών μειώθηκε κατά 30%. Από την άλλη πλευρά, μόνο 1% των ε, ιδιοκτητών μεγαλύτερης ηλικίας, 65 και άνω δηλαδή, μόνο 1,2 αποσύρθηκαν από την ε, παραγωγική διαδικασία. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα στοιχεία ήταν λίγο πιο θετικά, αλλά η μείωση μεταξύ των ηλικιωμένων, των πιο ηλικιωμένων ήταν πολύ λιγότερη από τη μείωση μεταξύ των νέων. Η διαφάνεια την οποία βλέπετε τώρα αναφέρεται στην τάση παραγωγών και την τάση, την πτωτική τάση στους αγρότες που είναι κάτω από 35 ή άνω των 65. Οι μπλε δείχνουν την μείωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αν μπορείτε να τη διακρίνετε την μπλε γραμμή, είναι η πτωτική τάση και η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κύπρο. Στην Κύπρο 60% μείωση μεταξύ των νέων παραγωγών, στην Εστονία 64, στη Ρουμανία 57. Το υπόλοιπο διάγραμμα αφορά άλλες χώρες και Βουλγαρία, Λιθωνία, Πορτογαλία και Ολλανδία έχουν ε, αρνητικές τάσεις, δηλαδή πτωτικές, πτωτικά στοιχεία. ενώ ελαχιστότατη αύξηση είχε η Σλοβενία, η Ελλάδα και η Τσεχία στον αριθμό των νέων. Αυτός ο χάρτης από τη Eurostat παρουσιάζει το μερίδιο των νέων παραγωγών κάτω από 35 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σκούρα χρώματα, τα κόκκινα και το πορτοκαλί ε, δείχνουν τους ε, καθαρούς αριθμούς, τα καθαρά στοιχεία, σε απόλυτα στοιχεία δηλαδή. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Το 2007 περίπου το 1 τρίτο των νέων παραγωγών ήταν ε, παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15, των 15. 33% λοιπόν είναι η παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες οι οποίες εντάξθηκαν το 2004 παρουσιάζουν 22% του μεριδίου των νέων παραγωγών και το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τις δύο νεότερες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία δηλαδή. Και αν θεωρήσουμε το μερίδιο, αν εξετάσουμε το συνολικό μερίδιο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θα δείτε ότι η χώρα μου, η Πολωνία, το 2007 είχε μια ικανοποιητική δομή 12,3% μερίδιο δηλαδή μεταξύ του συνολικού αριθμού των χρηστών 12,3% στην Πολωνία ήταν νέοι. Μετά έπεται η Τσεχία, Αυστρία, Φιλανδία. Από την άλλη πλευρά, στη δεξιά πλευρά έχουμε τα μικρά ποσοστά, τα μικρά μερίδια των νέων παραγωγών όπως η Πορτογαλία, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία. Οι νέοι ε, είχαν ένα πολύ μικρό μερίδιο στην Ιταλία κάτω από 3% όλων των αγροτικών μονάδων, ιδιοκτητών, ήταν νέοι. Εδώ παρουσιάζω τα ίδια στοιχεία βάση 2 ετών 2003-2007 βλέπετε τα ποσοστά λοιπόν το κόκκινο είναι τα στοιχεία του 2007 το κίτρινο 2003 βλέπετε λοιπόν ότι έχει μειωθεί σε πολλές χώρες ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών που κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, να είχαν συνταξιοδοτηθεί. Είναι σε συντάξιμη ηλικία. 65 και άνω. Στις περισσότερες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον για τους άνδρες, το συντάξιμο έτος ε, είναι 65. Βλέπουμε όμως ότι 4,5 εκατομμύρια γεωργοί αυτής της ηλικία όπου κανονικά θα έπρεπε να ζουν τη ζωή ενός συνταξιούχου έχουν ε, δραστηριοποιούνται σε παραγωγικές μονάδες. Και περίπου 400.000 είναι νέοι. Ορισμένες χώρες όπως Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ρωμανία, Ιταλία και η Λιθουανία το μερίδιο των ηλικιωμένων είναι 40% και. 65 Ένα πολύ μεγάλο λοιπόν μερίδιο των παραγωγών είναι άνω των 65 ετών σε αυτές τις χώρες. Και ο, το στοιχείο το οποίο πολλές φορές αναφέρεται όταν μιλάμε για ηλικιακέ ομάδες είναι κάτω των 35 και άνω των 65 ανά 100 παραγωγούς. Για κάθε 100 λοιπόν μονάδες ε, έχω τους δύο πίνακες για τις δύο ηλικιακέ ε, ομάδες. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι το εξής. Εάν το 2003 υπήρχαν αρκετές χώρες όπως η Γερμανία, η Φιλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία όπου αυτοί οι νέοι ε, ήταν περισσότεροι από τους άνω των 65 για κάθε 100 παραγωγούς ε, στη Γερμανία το 2003, για κάθε 100 είχαμε 204 νέους. Ναι, για κάθε 100, Ενώ τώρα, το 2007 η Γερμανία είναι δεύτερη. Ε, από 204 νέους πήγε στους 103 το 2007. Chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą bardzo często podkreśla się po to, żeby... Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία μείωση της συμμετοχής των νέων αγροτών από το 2003 στο 2007. Γιατί λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η πτωτική τάση, διότι οι νέοι παραγωγοί, οι νέοι αγρότες είναι σε πολύ δυσκολότερη θέση από ότι οι μεγαλύτεροι Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γη την οποία έχουν, όπου είναι οι διοκτήτες. Συνήθως στη Γερμανία οι παραγωγικές μονάδες τις οποίες λειτουργούν οι νέοι, εκμεταλλεύονται οι νέοι, είναι μεγαλύτερες από ότι αυτές τις οποίες εκμεταλλεύονται οι ηλικιωμένοι, οι μεγαλύτεροι, ενώ σε άλλες χώρες παρουσιάζεται το αντίθετο. Υπάρχει, διαπιστώνεται λοιπόν η τάση ότι Εάν οι νέοι κληρονομήσουν αγροτική γη, συνήθως εάν εκμετάλλευση είναι μεγάλη, ε, διατηρούν την μονάδα την παραγωγική και μένουν στο αγρο... στην ε, ε, παραγωγική διαδικασία. Εφόσον κληρονομήσουν λοιπόν μια μεγάλη εκμετάλλευση. Το άλλο στοιχείο που επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι η κρατική βοήθεια, η κρατική ενίσχυση και αυτή μπορεί να ε, ε, έχει επίπτωση στις, στις αναλογίες. Τώρα σχετικά με, τον, ε, με το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων όπου νέοι είναι ιδιοκτήτες, εδώ δεν συμφωνώ με ορισμένες εξέσεις που ε, συμπεραίνουν ότι συνήθως οι νέοι έχουν λιγότερη γη στη διάθεσή τους διότι δεν μπορούν να ε, επεκταθούν κλπ. Ε, το γεγονός είναι ότι σε ορισμένε χώρες οι νέοι αγρότες έχουν παραγωγικές μονάδες πολύ ψηλότερες από ότι ο μέσος όρος των εκμεταλλεύσεων και εάν θεωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 15, τα παλαιότερα μέλη, ο μέσος όρος μιας εκμετάλλευσης είναι 34 εκτάρια ενός νέου αγρότη, ενώ ο μέσος όρος σε όλη τη χώρα μεγέθους εκμετάλλευσης είναι 25 εκτάρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Δείχνει ακριβώς ότι πολλοί νέοι αγρότες έχουν μεγαλύτερες μονάδες. Στα καινούργια κράτη-μέλη η κατάσταση είναι αντίθετη, αντίστροφη. Αν ο μέσος όρος του κράτους μέλους είναι 22, οι νέοι ιδιοκτήτες θα είχαν γη μόνο 17 εκτάρια, 17 εκταρίων. Αντίστροφη. Δεν μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε. Ή οι μονάδες ε, οι οποίοι έχουν ιδιοκτήτες νέους αγρότες είναι σχετικά μεγάλες ή σχετικά μικρές και δεν μπορούμε να απαντήσουμε ξεκάθαρα με έναν ορισμό, με μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Έχουν οι νέοι μεγάλες ή μικρές εκμεταλλεύσεις σε ορισμένες χώρες όπως τη Δανία, την Εστονία, την Πορτογαλία. Οι μονάδες είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο, σε άλλες είναι μικρότερες. Η Εστονία είναι από τις χώρες, από τις νέες χώρες όπου οι εκμεταλλεύσεις είναι, αρκετά, είναι μεγάλες. Ε, και ενώ υπάρχουν παλαιά μέλη όπου οι νέοι έχουν μικρότερες εκμεταλλεύσεις στο Ενμένο Βασίλειο π.χ., στα παλαιά κράτη-μέλη, στη, στη Γερμανία. Επίσης, αλλά οι περισσότερες χώρες, οι περισσότερες από τις χώρες αυτές είναι καινούριε. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση των νέων παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και χρόνια έχουμε υλοποιήσει διάφορα προγράμματα ενίσχυσης όπως κρατική βοήθεια, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεση ή άμεση και πρέπει να ομολογήσω ότι παρόλο που ευρωβουλευτές των νέων χωρών πολλές φορές ισχυρίζονται ότι οι νέες χώρες υφίστανται αρνητική διάκριση Πρέπει ειλικρινά να πω ότι εάν δεν είχαμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νέοι μας αγρότες σε καμία περίπτωση δεν θα ελάμβαναν τόσες ενισχύσεις όπως λαμβάνουν τώρα. Βέβαια, όταν πάρεις κάτι, πάντα μεγαλώνει η όρεξή σου και θέλεις περισσότερο, διότι όπως λέμε το μάτι του ανθρώπου αχόρταγο. Και γι' αυτό ακριβώς καταλαβαίνω όταν ο κόσμος γκρινιάζει και παραπονιέται. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πώς βελτίωσε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δομές, τις αγροτικές ε, που, ενισχύουν τους νέους ε, παραγωγούς ή όσους έχουν υπόψη του να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Διότι από ό,τι κατάλαβα όταν μου δόθηκε η εντολή θα θέλατε να ακούσετε και ορισμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους αγρότες στον τομέα. Αυτό. Και να επιλέξουν αυτή τη σταδιοδρομία. Πρέπει να πω ότι εδώ έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα, διότι ακόμα και χτες με τους φοιτητέ μου ε, ε, ε, σε μια συζήτηση που κάναμε γενική ρώτησα τους φοιτητέ μου τους που προέρχονται από πόλεις, από αστικές περιοχές τι θα θέλατε να πάρετε, να κερδίσετε από το κράτος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα θέλατε, ποια κίνητα θα θέλατε για να μετακινηθείτε από αστικές περιοχές στην Ήπεθρο. Ορισμένοι γέλασαν ηρωνικά, αλλά ορισμένοι άλλοι φοιτητέ μου, μου είπαν τα εξή. Καταρχάς, κανένα χρηματικό ποσό δεν θα τους πείσει να μετακινηθούν από την πόλη στην Ήπεθρο. Διότι τους γιατί και μου είπαν ότι στην πόλη η ποιότητα της ζωής μου είναι υψηλή και Είμαι βέβαιος ότι στις αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθο και στα χωριά το επίπεδο τη ζωή μου θα μειωθεί, θα είναι πολύ χαμηλότερο. Διότι η αγροτική ζωή είναι σκληρή και η εργασία είναι σκληρή, έχει χειρονακτική εργασία και με κανένα, κανένα χρηματικό κίνητο δεν θα τους ε, έπεισε να μετακινηθούν από την πόλη στο χωριό. όταν τους ρώτησα τι εισόδημα θα θέλανε για να μετακινηθούν στην Ήπεθρο, οι απαντήσεις τους δεν ήταν ρεαλιστικές, διότι μου λέγανε ότι θέλουν ένα εισόδημα 150.000 σλότι το μήνα, ε, το οποίο είναι εκτός πραγματικότητος, δηλαδή να έχουν πενταπλάσιο μισθό του μέσου μισθού της Πολωνίας, των Πολωνών. Πενταπλάσιο μισθό για να πάνε στην επαρχία. Ε, άρα λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα σε αυτήν την μελέτη. Στην, ε, στην έκθεση αυτή και στην έκθεση του καθηγητή Σάξμις. Πιστεύουμε ότι τα χρηματικά κίνητρα, δάνεια, επιδοτήσεις κλπ. δεν πείθουν τους νέους. Για τους νέους η πρώτη προτεραιότητα είναι η ποιότητα της ζωής. Θέλουν να ζουν κοντά στους φίλους τους, να μην είναι απομονωμένοι, να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ιδέες τους, να έχουν ευελιξία στην καριέρα τους άλλοι παράγοντες δηλαδή πλην των καθαρών χρηματικών εισόδημα και κίνητρα οικονομικά. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθώ σε τρία προγράμματα τα οποία έχουν σχέση μεταξύ τους και με αυτό το, τη διαπίστωση. Το πρώτο πρόγραμμα του πρώτου άξονα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. για το ξεκίνημα μιας ε, αγροτικής ε, ή επιχειρησιακής ε, απασχόλησης στην Ήπεθρο. Είναι το μέτρο 112, δηλαδή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα και προώθηση κινήτρων και μέτρων όπως το 112 για, για το ξεκίνημα, την ε, δημιουργία νέων εκμεταλλεύσεων από νέους. Επίσης, ε, μέτρα προ πρόορης ε, συνταξιοδότησης το μέτρο 113. Πιστεύουμε ότι στην Πολωνία ε, είχαμε πολύ χαμηλά πριν, περίπου 50.000 πολωνικά σλότη ε, για την ενίσχυση των αγροτών και σε άλλες χώρες αυτή η ενίσχυση ήταν πολύ μεγαλύτερη αλλά φέτος αυξήθηκε κατά 50% και Έχουμε επίσης, εκτός από αυτές τις ενισχύσεις, όπως είπα, και κίνητρα για την πρόορη συνταξιοδότηση. Ίσως μπορούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα συνδυασμό τέτοιων ε, μέτρων. Δηλαδή να μην ενισχύσουμε μόνο την πρόορη συνταξιοδότηση, αλλά να συνδυάσουμε επιδότηση για την ε, ε, κίνηση μιας αγροτικής μονάδας, ε, ε, ε, πρόορη συνταξιοδότηση και επαγγελματική κατάρτιση και δραστηριότητες πληροφόρησης. Μέτρο 111. Η δράση 111. Αυτές οι τρεις δράσεις 112, 113, 111, 1-13, μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω. Για πολλούς ανθρώπους λοιπόν όπως σας είπα προτεραιότητα δεν έχει η αγροτική παραγωγή αλλά η διατήρηση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τους ενδιαφέρει σαφώς η ποιότητα της ζωής τους. Γι' αυτό πρέπει να βελτιωθεί στην Ήπεθρο η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων ε, ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ αστικών και αγροτικών ε, περιοχών. Ε, Πολλοί θα ήθελαν να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν μια καλή ποιότητα ζωής. Οι, άνθρωποι που, οι νέοι άνθρωποι ζητούν πολλά, ζητούν περισσότερα. Ένα άλλο στοιχείο είναι η προσφορά βασικών υπηρεσιών. Σήμερα το πρόβλημα των νέων ανθρώπων στην Ήπεθρο είναι ότι υποφέρουν από νοητικές ασθένειες, παραδείγματο χάρη κατάθλιψη. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από την Κοινοβούλιο και την Κομισιόν ε, να, να τους ρωτήσω εάν έχουν κάνει μία, ένα τσεκ υγείας της κοινή αγροτικής πολιτικής, αν μπορούν να κάνουν και ένα τσεκ υγείας ε, ε, της, των νέων γεωργών. Ε, γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις βασικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας. Ε, οι βασικές υπηρεσίες βεβαίως καλύπτουν όχι μόνο τους νέους γεωργούς αλλά όλο τον πληθυσμό. Αν θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι να ζουν εκτός πόλεων πρέπει να βελτιώσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και ο τέταρτος άξονας ε, είναι το leader Α, είναι η ανάπτυξη ηγετικών προσόντων, δηλαδή να μπορεί κάποιος να οργανώσει μια τοπική ομάδα δράσης, να αναλάβει πρωτοβουλίες κλπ. Θέλουμε περισσότερες ε, αρχηγικές ε, φυσιογνωμίες, αρχηγικές προσωπικότητες. Και έχουμε το Συμβούλιο των Νέων Αγροτών και πολλούς φορείς τέτοιους και κάποιος πρέπει να λάβει την ηγεσία τους. Οι πολλοί νέοι αγρότες μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει αρκετή προσοχή σε νέους παραγωγούς. Εάν όμως όλα αυτά τα ε, ε, προγράμματα ε, έχουν καλύπτουν μόνο νέους γεωργούς τότε θα μείνουν εκτός ενίσχυσης πολλά άλλα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, υπήρχε ιδέα ενό προγράμματο ε, για την βελτίωση ε, των συνθηκών εγκατάσταση νέων αγροτών, αλλά ούτε καν ξεκίνησε ε, σε πολλέ από τι νέε χώρε, όπω τη Σλοβακία. Και σε πολλές ε, περιφέρειες της Γερμανίας το, τα προγράμματα αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Παραδείγματο χάρη στην Ουαλία καθόλου δεν προχώρησε αυτό το θέμα, αλλά στην Ιρλανδία και, σε ορισμένε χώρε όπω την Ιρλανδία που ξεκίνησε αυτό το μέτρο βοήθεια, α πούμε, εν συνεχεία καταργήθηκε. Λόγω της οικονομικής ε, Στις τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές αυτό το μέτρο δεν έχει καθόλου περιληφθεί στις 17 ε, ε, χώρες, σε 17 χώρες και μπορείτε να δείτε τον κατάλογο αυτών των χωρών. Όμως όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τις ε, ενέργειες δράσης ενημέρωσης μέτρο 111 έχουν ξεκινήσει ορισμένα προγράμματα σε περιφέρειες ε, ε, των κρατών μελών σε άλλες περιφέρειες όμως όχι όπως ε, σε ορισμένα κρατήδια της Γερμανίας εδώ έχω, έχω διαφορετικά αποκλίνουσες πληροφορίες ότι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το 3,3% των προγραμμάτων υπό τον πρώτο άξονα έχουν ξεκινήσει. αυτή η διαφάνεια πάλι εδώ μας δείχνει την κατανομή των πιστώσεων για νέους αγρότες. Μόνο 10% του πρώτου άξονα υπό τον πρώτο πυλώνα και 3% ε, στο δεύτερο πυλώνα ή αντίστροφα. Ε, δεν, ε, βλέπετε τον πίνακα πάντως. Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις θα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω και τώρα θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε νέους παραγωγούς στον τομέα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως ε, στελέχη που αποφασίζουμε για την πολιτική. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλους ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου και αυτούς που ασκούν πίεση, τους λόμπιστ, ε, γιατί θέλουμε σε πολλές, αν όχι σε όλες χώρες, να υπάρξουν τα μέσα αυτά, γιατί συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του, της κατανομής του πληθυσμού, στην Ήπεθρο. Τα προγράμματα προγράμματα και τα μέσα αυτά ε, πολύ συχνά βοηθούν τους νέους να στραφούν στη γεωργία. Επειδή για το θέμα συζητούμε τόσο πολύ, θα ήθελα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Αν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να προτείνουμε νέα μέσα. Στην έκθεσή μου ε, ε, τα χώρισα τα εμπόδια σε ομάδες Θέλω λοιπόν να προτείνω μια ιδέα που αφορά σε γενικές λύσεις. Δεν είμαι πάρα πολύ έμπειρη σε αυτό το τομέα, δεν είμαι πολιτικός, ο τομέας είναι εξαιρετικά εκτεταμένος, τα πάντα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της μελέτης επιπτώσεων και μια σειρά από άλλα. Έτσι λοιπόν μερικές πρώτες ιδέες. Το πρώτο εμπόδιο το οποίο πολύ συχνά το αναφέρουν οι ίδιοι οι νέοι και οι οργανισμοί τους είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στα κεφάλαια. Ε, επίσης πώς θα βρεθεί μια καλή γη. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να την κληρονομήσει κανείς. Όμως αυτό δεν είναι πολύ ε, ε, συνηθισμένο. Αυτό το παλιό μοντέλο της κληροδότησης της γης από τη μια γενιά στην άλλη ε, δεν υπάρχει παντού στην Πολωνία. Στην Ελλάδα υπάρχει αλλά όχι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν και χώρες όπως η Πολωνία και η Ελλάδα που έχουν και αυτές προβλήματα γιατί πολλοί γονείς δεν έχουν παιδιά και δεν θέλουν να μεταβιβάσουν τη γη τους σε ξένους και πολύ συχνά ε, διατηρούν τη γη εν είδη κεφαλαίου και ο κόσμος περιμένει ότι θα ανεβεί η τιμή της γης και ίσως η, η γη αυτή να ε, ε, να αλλάξει χρήση, ε, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν, να κάνουν τη γη τους οικόπεδα κλπ. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Προσπάθησα να πάρω στοιχεία από την Eurostat και, από, και να στραφώ σε διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων. Δεν υπάρχουν όμως στατιστικά στοιχεία που να λένε πόσα άτομα στα κράτη-μέλη ή και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν μια αγροτική δραστηριότητα. Και επίσης δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για το πόσοι νέοι το χρόνο κληρονομούν γη από τους γονείς τους ή στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα στοιχεία δεν μπόρεσα να τα βρω. Στις χώρες λοιπόν αυτές οι οποίες ε, υπάρχει παραδοσιακή μορφή, μορφή γεωργίας, οικογενειακή γεωργία. Ε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τους γονείς να τους αγρότες μάλλον να μεταβιβάζουν τη γη τους σε ξένους πρέπει να δώσουμε πολύ ισχυρά κίνητρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μεταβιβάσουν τη γη τους σε, ανθρώπους που τους είναι παντελώς άγνωστοι. Ε, ξέρω ότι αυτό ισχύει στην Πολωνία αλλά και ίσως και σε άλλα κράτη-μέλη ότι υπάρχουν χώρες που ενδιαφέρονται να ε, δώσουν μια συνέχεια ε, στα προγράμματα είτε της ε, πρώιμης χρηματοδότησης είτε της ενίσχυσης ε, του ξεκινήματος δραστηριότητας σε αυτούς τους τομείς. Σε κάποιες χώρες ίσως να μην χρειάζεται συνδυασμό αυτών των δύο μέσων, ίσως να μην χρειάζεται η πρώιμη, χρηματοδο... συνταξιοδότηση, αλλά σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ελλάδα, για, τι για τις αυτές θα πρέπει το να εισαχθούν αυτά τα προγράμματα, να υλοποιηθούν, αλλά από κοινού. Και υπάρχει και μια άλλη ιδέα που αφορά τη προγράμματα δημιουργίας και ανάπτυξης ε, και που στοχεύουν στους ε, ε, μεγαλύτερης ηλικία αγρότες. Να είναι προγράμματα αποταμίευσης μεγαλύτερων σε ηλικία αγροτών με αυτόν τον τρόπο ίσως αυτοί οι άνθρωποι ε, βοηθηθούν να συγκεντρώσουν ε, κάποιο κεφάλαιο για μια μετέπειτα φάση της ζωής τους. Και μπορεί κανείς να υποθέσει ότι από τη στιγμή που θα έχουν κάποιες αποταμιεύσεις, κάποιες οικονομίες και αν τους δοθεί και κάποια πρώτη μισιακή μεταχείριση για τις οικονομίες τους αυτές, τότε αν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ε, μεταβιβάσουν τη γη τους σε μια ηλικία άνω των 50 ετών, ε, να έχουν τις οικονομίες τους υπό την προϋπόθεση είπαμε ότι θα μεταβιβάσουν τη γη τους. Στα άλλα κράτη-μέλη το κόστος αυτής της συναλλαγής είναι πάρα πολύ ψηλό. Ε, τα συμβολιογραφικά έξοδα λοιπόν, ε, ο έλεγχος των εγγράφων και η όλη γραφειοκρατία συνεπάγονται πολύ ψηλό κόστος που καμιά φορά συνοδεύεται και από δίκες λόγω λαθών κλπ. Θα ήταν λοιπόν εδώ κάποια βοήθεια χρήσιμη, ίσως, ίσως ευρω... όχι ίσως ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κάποια στήριξη κάποιο, ε, αυτού του, του κόστους. Ένα άλλο πολύ συχνό εμπόδιο είναι η έλλειψη πρόσβασης στο ε, κεφάλαιο, σε κεφάλαια. Είμαι οικονομολόγος και κάπως φιλελεύθερη. Αν ε, έλεγα ε, αυτά που πιστεύω για τις δημόσιες ενισχύσεις, νομίζω ότι πολλοί θα διαφωνήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είχα εγώ να επιλέξω ανάμεσα σε ε, επιλογή τέτοιων πληρωμών, τέτοιων καταβολών και δάνειων, πιστεύω ότι αυτές οι πληρωμές είναι προτιμότερες. Γιατί αν κανείς πάρει μια πίστοση, ένα δάνειο, πρέπει να αποπληρωθεί αυτό. Αυτό απαιτεί από τους ε, ε, χρηματοδοτούμενους μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αν όμως πάρω δωρεάν ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν προσέχει πώς θα δαπανίσω τα λεφτά μου και πάρα πολύ συχνά τα χρήματα αυτά χάνονται, σπαταλώνται, ενώ το δάνειο πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ε, ορθολογικό. Φυσικά ε, το θέμα αυτό είναι της εθνικής αρμοδιότητας, θα μπορούσαν να δοθούν ε, κάποιες, κάποιοι προτιμησιακοί όροι. Υπάρχει η βοήθεια ντεμίνιμης, η ενίσχυση ντεμίνιμης που ε, τα δάνεια με προτιμήσιακού όρους σε νέους αγρότες. Όμως αυτή του είδου η χρηματοδότηση δεν είναι εύκολη. Τα κριτήρια και οι προποθέσει είναι πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω με τι λεπτομέρειες. Πάντως ε, είναι πολλά τα προαπαιτούμενα. Εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε ίσως να δημιουργήσουμε κάτι, ίσως όχι μια ακόμα τράπεζα, αλλά ένα είδος προγράμματος στήριξης. Ένα πρόγραμμα που να προσφέρει κεφάλαιο ή δάνεια. Έχω κάποιους φοιτητές που έχουν προτείνει κάποια λύση ένα μεγάλο κεφάλαιο που να προέρχεται από φόρους ή άλλες πηγές και ε, το θεσμικό όργανο που κατέχει το κεφάλαιο και που ενδεχομένως γνωρίζει τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους ε, θα μπορούσε να δανειοδοτεί κράτη-μέλη και κατόπιν τα κράτη-μέλη να κάνουν την κατανομή ε, των χρημάτων. Βεβαίως ε, εδώ και εδώ θα πρέπει να ισχύουν κανόνες. Αν ένας νέος αγρότης δανειοδοτηθεί ή αν ένας ε, ε, κάποιος που θέλει να γίνει νέος αγρότης δανειοδοτηθεί και τελικά εγκαταλείψει τη γεωργία τότε θα πρέπει να επιστρέψει ε, τα χρήματα. Να υπάρχει δηλαδή και κάποιο σύστημα ποινών. Ε, κύριε Πρόεδρε έχω λίγο χρόνο παραπάνω. Ωραία. Οπότε μπορώ και να συνεχίσω. Τέσσερις χώρες ε, Ανατολικής, για τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης έχουμε το πρόβλημα της πρόσβασης στον εξοπλισμό, στα εργαλεία. Στην Πολωνία υπήρχε ένα σύστημα ε, συνεταιρισμών όπως τους αποκαλούσαμε. Ε, όπου μπορούσε κανείς να νοικιάσει τον εξοπλισμό ως αγρότης αν δεν μπορούσε να τον αγοράσει. Πολύ συχνά οι νέοι αγρότες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να αγοράσουν όλο τον εξοπλισμό που τους χρειάζεται και χρειάζεται να προχωρήσουν σε χρονομίσθωση για, ή να δανειστούν για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό. Πρέπει να προσφέρουμε κάποιο είδους στήριξη σε αυτούς τους συνεταιρισμούς οι οποίοι ε, προσφέρουν ε, ε, με τρόπο οικονομικό εξοπλισμό στους νέους αγρότες. Επίσης υπάρχει ένας κίνδυνος. Ε, διέτρεξα τα φόρουμ συζητήσεων που υπάρχουν στην αγγλική γλώσσα για τους νέους. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ε, όλες αυτές οι ιστοσελίδες που αφορούν τους νέους αγρότες δεν είναι όλες στα αγγλικά. Φοβάμαι ότι όλες αυτές οι πληροφορίες ε, που υπάρχουν στο διαδίκτυο θα πρέπει να υπάρχουν στα αγγλικά γιατί αλλιώς δεν, μπορούμε, δεν θα μπορέσουμε να τις αναλύσουμε. Εν πάση περιπτώσει διέτρεξα όλους τους χώρους ε, συζήτησης και διαπίστωσα ότι πολύ συχνά οι νέοι λένε ναι υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει ένα εμπόδιο που τους εμποδίζει από το να ασχοληθούν με την γεωργία. Ο κίνδυνος ε, πράγματι, εδώ υπάρχουν προβλήματα. Στην ε, Πολωνία, ας πούμε, είχαμε πλημμύρες, ξηρασία τα Ε, γι' αυτό αυτό ίσως να φοβίζει τους νέους. Επίσης, ε, μελέτησα τα ασφαλιστικά προγράμματα στα κράτη-μέλη ε, ασφάλειες της αγροτικής παραγωγής και βρήκα ότι μόνο στην Ισπανία και στη Γαλλία υπάρχουν Εκεί δίνεται κάποια προτιμησιακή μεταχείριση στους νέους αγρότες όσον αφορά την ασφάλιση. Δηλαδή, το 50% το κατέβαλε ο αγρότης και το 50% το συγχρηματοδοτούσαν οι αρχές. Μόνο όμως σε δύο κράτη-μέλη το βρήκα αυτό. Δεν μπόρεσα να βρω κανένα άλλο κράτος μέλος στα οποίο να προσφέρεται προτιμησιακή μεταχείριση ε, ασφαλιστικής πολιτικής ε, στους νέους αγρότες. Γνωρίζω βεβαίως ότι η ΚΑΠ δεν καλύπτει τα, ε, τα θέματα ασφάλισης πρέπει να συνεχίσουμε ε, να στηρίζουμε τις εθνικές κυβερνήσεις, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να ε, αναγκαστούν να συμπεριλάβουν και αυτό το θέμα της ε, ασφαλιστικής κάλυψης των νέων αγροτών. Ε, οι φοιτητέ καμιά φορά προτείνουν απλέ λύσει. Λένε α πούμε πρέπει να, δίνεται, να χορηγείται μια περίοδο χάριτος στην ασφάλιση και στα δάνεια. Πρέπει στου νέου αγρότε να χορηγείται μια μακρύτερη περίοδο χάριτος για να του διευκολυνθούν. Ή σε αναδυόμενου κλάδου δίνεται αυτό. Οι νέοι αγρότε είναι και αυτοί ένα αναδυόμενο χώρο. Πρέπει λοιπόν να στηρίζονται περίοδο χάριτος, να του δίνεται από τι τράπεζε κτλ. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι αγρότες ζουν στην Ήπεθρο. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στην Ήπεθρο ε, έχουν στόχο και τους νέους αγρότες. Όμως οι νέοι αγρότες είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι. Θέλουν να βγαίνουν, να πάνε σινεμά, στο θέατρο, να πάνε να πιούν. Ε, σε αυτές, στην Ήπεθρο δεν υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές. Χρειάζονται λοιπόν καλύτερες υποδομές. Ίσως να υπάρχουν δρόμοι, αλλά δεν υπάρχουν λεωφορεία, μέσα μεταφοράς ή χώροι ψυχαγωγίας. Ε, πολύ συχνά... Ε, ε μας απαντούν πάρτε ε, κι άλλο αυτοκίνητο. Ναι, αλλά τι θα γίνει, κάθε οικογένεια θα έχει τέσσερα αυτοκίνητα, αυτό κοστίζει πολύ. Επίσης, ε, και αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αν όμως να δαπανηθούν χρήματα για την κατασκευή δρόμων, πρέπει να δοθούν χρήματα για να στηριχθούν οι τοπικές αρχές, να μπορούν ας πούμε, να καλύψουν το κόστος χρηματοδότησης μέσων ε, μεταφοράς μεταξύ του χωριού ας πούμε και μιας μεγαλύτερης πόλης. Και εγώ στην Ήπεθρο ζω Ε, οι γονεί μου κατοικούν και αυτοί σε μια περιοχή της Πολωνίας και όταν ήμουν φοιτήτρια υπήρχαν 5-6 λεωφορεία κάθε μέρα για την περιοχή. Αλλά τώρα, από ό,τι ξέρω, μόνο μόνο ή 3 λεωφορεία υπάρχουν και το καλοκαίρι ακόμα λιγότερα. λιγότερα. Ε, 2-3 λεωφορεία που να συνδέουν ε, την Ήπεθρο με την πόλη. Ο κόσμος λοιπόν ε, δεν μπορεί να ξεφύγει από την Ήπεθρο. Υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς. Δεν έχουν τα μέσον, έχουν τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να ε, ψυχαγωγηθούν. Επίσης υπάρχει το θέμα της υγείας των νεαρών αγροτών. Ε, οι έρευνες που έγιναν στη Βρετανία διαπιστώνουν ότι οι νέοι αγρότες είναι πιο ανθεκτικοί σε κάποιες ασθένειες και παθήσεις. Βεβαίως υπάρχει πάντα το θέμα των ατυχημάτων ή υπάρχουν οι, οι ασθένειες που προκαλούνται από τη χρήση των λιπασμάτων. Υπάρχει όμως και το θέμα της ψυχικής ασθένειας. Υπάρχει ε, τεράστιο άγχος, στρες ε, που έχει σχέση με το κίνδυνο, με, τις, με το οικονομικά. Τελικά εδώ μιλάμε για προσέλκυση νέων στον κλάδο αυτό. Οι δυσκολίες είναι πολλές. Το θέμα το έθιξε και ο καθηγητής που ε, αναφέρθηκε ε, στην, στα θέματα της εκπαίδευσης. Και πρέπει να πω ότι δεν μιλάμε τώρα μόνο για το γεγονός ότι είναι πολύ λίγοι οι αγρότες που έχουν πτυχίο της εκπαιδείας. Ε, έχω τα στοιχεία του 2005 που δείχνουν ότι ε, μόνο το 20% των ε, αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποιο είδους αγροτική κατάρτιση. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Στη Μάλτη είναι κάτω από το 1% αυτό το ποσοστό ε, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στη Μάλτα ε, γιατί το πρόγραμμα ε, που ενισχύει την δραστηριότητα εκκίνησης έχει κάποιες προϋποθέσεις. Οι καλύτερα, οι περισσότερο μορφωμένοι αγρότες βρίσκονται στις κάτω χώρες και τη Γερμανία. Όταν όμως συζήτησα με τους φοιτητές μου για το θέμα αυτό, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Αυτοί που ε, έχουν σκοπό να επιστρέψουν στην Ήπεθρο λένε ότι η εκπαίδευση, η μόρφωση είναι σημαντική γιατί τη σήμερα μέρα πρέπει κανείς να μπορεί να κάνει ε, να τηρήσει λογιστικά βιβλία, να μπορεί να συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα business plan, να γνωρίζει τη χρήση του υπολογιστή. Δηλαδή δεν απαιτείται μόνο η γνώση για την αγροτική παραγωγή, αλλά γενικές γνώσεις. Και πολύ συχνά οι νέοι αγρότες παραπονούνται ότι δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και γι' αυτό υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Φερρυπίν δεν είναι εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο. Κυρίως όμως αυτό αφορά τον τρόπο και την μέθοδο διάδοσης των πληροφοριών. Ενδεχομένως θα μάθατε τα αποτελέσματα του πρόσφατου ευρωβαρομέτρου που αφορά ε, την ε, αγροτική πολιτική των ε, κρατών μελών. Έφρυξα η λέει, αναφέρει ότι αν το 50% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακούσει ποτέ τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική. μόνο φρίκι μπορεί να μου προκαλέσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα το 50% των ανθρώπων δεν έχουν ακούσει ποτέ για την ΚΑΠ την ώρα που τόσα δαπανώνται για αυτήν. Έχουν γίνει λοιπόν έρευνες τις οποίες δεν διαβάζει κανένας. Θα έπρεπε πιστεύω να γίνει κάποια ενημερωτική εκστρατεία από τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο για να ενημερωθεί ο κόσμος τι ακριβώς είναι η κοινή αγροτική πολιτική. πιστεύω ότι πρέπει να ε, ενημερώσουμε τους πολίτες μας ποιοι είναι οι αγρότες και τι σημαίνει αγροτική παραγωγή. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, εκ των κάτω προς τα άνω. Οι δικοί μου φοιτητές πολύ συχνά όταν τους ρωτάω ε, αν ε, έχουν περάσει από κάποια επαγγελματική κατάρτιση πριν επιλέξουν την σχολή στην οποία πηγαίνουν, μου λένε όχι δεν ε, έχουν περάσει από κανέναν επαγγελματικό προσανατολισμό, ποτέ δεν τους εξήγησαν τι ευκαιρίες υπάρχουν, τι επαγγελματικές δυνατότητες υπάρχουν, κανείς δεν τους μίλησε για τα υπέρ και τα κατά κάποιου ε, επαγγέλματο. Θεωρούν ε, μάλιστα οι φοιτητέ μου ότι πρέπει πολύ νωρί να γίνεται αυτού του είδου ο επαγγελματικό προσανατολισμό, ήδη από το δημοτικό σχολείο να αρχίσουν οι άνθρωποι να ενημερώνονται για τι επιλογέ του οι νεαροί αγρότες πολύ συχνά υποτιμώνται, διότι υπάρχουν και αυτοί που έχουν μεγάλη επιτυχία. Ε, έχουμε στην Πολωνία νεαρούς αγρότες που είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι, ε, παιδιά που είναι ενήμερα, ε, που έχουν πολύ σύγχρονες μονάδες, αλλά δεν είναι γνωστοί. Γίνεται μια εκπομπή για την Ήπεθρο ε, στην Πολωνία την Κυριακή, αλλά ποιος τη βλέπει αυτή στις 12 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής. Υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες αγρότες. Ε, τέλος, ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερο λόγο οι αγρότες, οι νέοι αγρότες. Θα πρέπει να τους ρωτάμε και να ακούμε τους νέους γενικά στα σχολεία, να ακούμε τις προτιμήσεις τους, να συζητάμε ε, για την ύπεθρο, για τις αγροτικές περιοχές και όταν η προσέγγιση τους είναι αρνητική να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Îi Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία μου για αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο κύριος Μπέκερ, πρόεδρος του ΣΕΖΑ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μόνιμων αντιπροσωπιών, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπέθρου, τον Παύλο Ντεκάστρο, που ο οποίος ε, οργάνωσε και έδωσε τη δυνατότητα να ε, πραγματοποιηθεί σήμερα εδώ αυτή η ημερίδα. Στην πραγματικότητα πάρα πολλοί νέοι αγρότες παρίστανται σήμερα το απόγευμα για να παρακολουθήσουν τις εργασίες. Οι συναντήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικές για μας. Είμαστε σε τακτική επαφή μαζί σας. Ε, είναι πρόσδεκτη αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα, η οποία, ε, χάρη στην οποία προσκλήθηκαν δύο εμπειρογνώμονες ε, για να συζητήσουν την κατάσταση των νεαρών αγροτών και της νεολαίας Τη υπαίθρου στην Ευρώπη. Η κυρία Ζαβόσκα επεσήμανε διάφορα θέματα και που απασχολούν τους νέους αγρότες όπως επίσης και τις διαφορές στην εφαρμογή ε, των μέτρων για τους νέους αγρότες στην Ευρώπη. Εμείς η ΣΕΖΑ ε, είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε πίσω από όλα τα νούμερα που αναφέρατε σήμερα. Ε, οι νεαροί άνδρες και γυναίκες ενδιαφέρονται να μπουν στην αγροτική παραγωγή. Οι άνθρωποι που έχουν μόλις μπει και προσπαθούν να, να προχωρήσουν ε, ως νεαροί ε, επιχειρηματίες του αγροτικού χώρου. Ε, οι οποίοι θέλουν να παράγουν τις τα υψηλής ποιότητας τρόφιμα και δημόσια αγαθά που θα χρειαστεί τώρα και στο μέλλον η ευρωπαϊκή κοινωνία. Βρισκόμαστε εδώ για να σας ζητήσουμε να μας στηρίξετε και να δημιουργήσουμε μια νέα κάπη η οποία να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των νεαρών αγροτών έτσι όλες, όλες οι προσδοκίες ε, ε, που έχει η κοινωνία από τη Γεωργία να υλοποιηθούν. Χτες και σήμερα οι νεαροί αγρότες από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ε, ποιε είναι οι σκέψει μα σχετικά με τη βελτίωση του μέλλοντο. Θα σα πω ποιε είναι οι σκέψει μα. Οι νέοι αγρότε μπορούν να σημειώσουν ότι αυτή τη στιγμή η ανανέωση των γενεών δεν θεωρείται ε, προτεραιότητα από πάρα πολλά κράτη-μέλη. Τα στοιχεία όπω τα παρουσίασε και η κυρία Ζαβόσκα είναι ξεκάθαρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών συνολικά μόνο το 3% των προγραμματισμένων δημοσίων δαπανών για τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ για το διάστημα 2007-2013, δηλαδή συνολικά 10% της ε, ε, συνολικής δημόσιας στήριξης που παρέχεται υπό τον άξονα 1 δαπανήθηκε στο μέτρο 112, μόνο το 10%. Λοιπόν, ζητώ από εσά τους ευρωβουλευτές να στηρίξετε την έκκληση των νέων αγροτών για να αλλάξει αυτή η τάση. Αν θέλουμε να παρέχει η γεωργία, διατροφική ασφάλεια, περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως επίσης και μια εδαφική ισορροπία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε νέους καινοτόμους και ε, επιχειρηματίες, ε, ε, νέους αγρότες που να είναι δυναμικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι φιλόδοξη στους στόχους της και να εγκαταστήσει τους νέους ερχόμενους και τους νέους αγρότες οι οποίοι συνεισφέρουν στους στόχους που ανέφερα παραπάνω και στη δημιουργία και τη συντήρηση απασχόλησης και θέσεων εργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά που υπάρχουν υπό τον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει και να ενισχυθούν και να αλλάξει μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ζητάμε ότι η βοήθεια στην εγκατάσταση, η ενίσχυση στην εγκατάσταση να είναι διαθέσιμη σε όλους τους νέους αγρότες και τους νέους ερχόμενους στον κλάδο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή κάποια κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν την ενίσχυση εγκατάστασης που διατίθεται από το δεύτερο πυλώνα. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισοτιμία όσον αφορά τους νέους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μία, ένα, μία αναθεώρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης χρηματοδότησης πρέπει να γίνει δεχτή ώστε να δοθεί πραγματικό κίνητρο και ευκαιρία στα κράτη-μέλη να θέσουν προτεραιότητα, την, ως προτεραιότητα την ε, ανανέωση των γενναιών. δηλαδή ένα ποσοστό 80 ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 20 εθνική χρηματοδότηση θα πρέπει να αντικαταστήσει το ισχύον 50-50. Επιπλέον το ανώτατο ποσό για την, ενίσχυση εγκατάσταση θα πρέπει να σταματήσει. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, το ποσό της εγκατάστασης έχει ανώτατο όριο. Αυτό είναι μια παράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει το ποσό της ενίσχυσης να είναι διαθέσιμο σε όλους και στα παλαιά και στα νέα κράτη-μέλη. Επίσης ζητάμε για έναν ισχυρό προπολογισμό που σύμφωνα με τη νέα ε, κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι ε, διαθέσιμος για τα μέτρα που στοχεύουν στην ανανέωση των γενεών και την είσοδο ομάδων νέων ε, αγροτών στον κλάδο. Ε, ο πρώτος ε, στον πρώτο πυλώνα ε, η ΣΕΖΑ ζητά ε, ένα συμπληρωματικό ε, πριμ για τους νέους αγρότες όπως επίσης και τη δημιουργία ενός αποθεματικού για τα ταμεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να ξαναδαπανηθούν στους νέους αγρότες. Η ΣΕΖΑ επίσης ζητά την ενίσχυση των μέτρων που στηρίζουν τα, τις επενδύσεις για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία πυρήνων. Στην πράξη η ενίσχυση εγκατάστασης θα πρέπει να να περιλαμβάνει και μια προτιμησιακή πρόσβαση για τους νέους αγρότες στα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σύμφωνα ε, στο, χώρο της αγροτικής ανάπτυξης. Τα επιδοτούμενα δάνεια θα πρέπει να συνδέονται με τις επενδύσεις που κάνουν οι νέοι αγρότες και θα πρέπει να διατίθενται όταν ε, οι νέοι αγρότες θέλουν να συνεργάζονται, να φτιάχνουν ε, συνεταιρισμούς ή συνεργασίες και δίκτυα η πολιτική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη για τη στήριξη της ανανέωσης των γενναιών στην οντομία της γεωργίας. Θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει και τα κουπόνια γνώσης ε, που θα χρησιμοποιούν οι νέοι αγρότες. Αυτά τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε, ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση σε νέες μεθόδους παραγωγής, η διαφοροποίηση των μονάδων, η φυτογειονομική εκπαίδευση, απευθείας πώληση, μάρκετινγκ κτλ. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζονται μόλις κάποιο ποσοστό ετοιμάτων από νέους αγρότες έχει καταγραφεί. Το πακέτο των νέων αγροτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, εκπαίδευση των νέων αγροτών στο εξωτερικό, όπως είπε και η κυρία Ζεβόσκα. Ένα είδος εράσμους για νέους αγρότες που θα ε, το παρακολουθούν ακριβώς πριν αναλάβουν την επιχείρηση αναφερθήκαμε προηγουμένως και στο πρόγραμμα ε, χρηματοδότησης ε, που θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της ΚΑΠ γιατί έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά του. Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι η ΣΕΖΑ χαιρετίζει την κατεύθυνση που προτείνει η Κομισιόν για τους ενεργούς αγρότες. Πριν από δύο εβδομάδες παρακολούθησα εδώ μια συζήτηση ευρωβουλευτών οι οποίοι αντιδρούσαν στην ανακοίνωση των ε, επιτρόπων για το μέλλον της ΚΑΠ. Πολλοί από εσά ε, έβαλαν ερωτήσεις για τους ενεργούς αγρότες. Θέλω να επαναλάβω ότι για μας είναι ακριβώς η σωστή κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΚΑΠ στο μέλλον. Δηλαδή, οι ενεργοί αγρότες για μας είναι αυτοί οι οποίοι ε, αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη διαχείρισης της επιχείρησης και της παραγωγής, οι οποίοι πουλάνε προϊόντα ατομικά ή μέσω συνεταιρισμών. Είναι επίσης αυτοί που τους αναγνωρίζει η δημόσια διοίκηση και είναι επίσης αυτοί οι οποίοι παραδίδουν ε, αγαθά λόγω, προερχόμενα από την αγροτική τους δραστηριότητα. Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι εμείς στη ΣΕΖΑ παρακολουθούμε το έργο σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από, ε, από κοντά. Ε, θα γνωρίζετε ότι πριν από ε, μερικά χρόνια η Κομ Άγκρη έγραψε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για την κατάσταση των νέων αγροτών. Τώρα όπου βρισκόμαστε στη διαδικασία μιας νέας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ ελπίζουμε ότι η νέα αυτή η Κομ Άγκρη που έχει αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να συνεχίσει να, δίνει, ε, ε, να στοχεύει στους νεαρούς αγρότες μετά από, αυτό το, από αυτή την ημερίδα. Μια έκθεση για τη συγκεκριμένη κατάσταση των νέων αγροτών θα είναι πρόσδεκτη. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να προσκαλέσω όλους σας σε μια εκδήλωση ε, στις 15 Δεκεμβρίου. Ο τίτλος είναι «Η επένδυση στις ε, ευκαιρίες των νέων αγροτών σε μια πολυλειτουργική γεωργία». Θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου, όπως σας είπα, στις Βρυξέλλες, στο κτίριο της ΟΚΕ και όλοι σας θα λάβετε ξεχωριστή πρόσκληση. Εν κατακλείδη, κύριε Ντεκάστρο, για μία ακόμα φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας προσφέρατε να συζητήσουμε σήμερα σε βάθος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι νέοι αγρότες και οι νέοι εισερχόμενοι στον κλάδο, όπως επίσης και τις λύσεις για τη διατήρηση και στήριξη μιας δυναμικής επιχειρηματικής και γεωργίας η οποία να βλέπει προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της ΣΕΖΑ. ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε σε όλα αυτά, γι' αυτό θελήσαμε να οργανώσουμε αυτό το εργαστήριο στους νέους και στην κοινοτική πολιτική που έχει να κάνει με τους νέους γεωργούς. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε, όπως επίσης την κυρία Ζαρβόσκα για όσα είπε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει η συζήτηση τώρα και στη συνέχεια θα λάβει την λόγο η Επιτροπή. Ξεκινάει η συζήτηση με τον κύριο Ταραμπέλα. Ο Μάρκ Ταραμπέλα έχει το λόγο. Αντιμετωπίζουμε κάποια προβληματάκια με τα μικρόφωνα σήμερα, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε κάποιο που να δουλεύει.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τα, τους δύο εισηγητές μας και για ορισμένου αριθμούς μας τρομάζουν αυτά, αυτά που είπε η κυρία στο ξεκίνημα της εισήγησής της. Το πόσο όλα αυτά χαλάνε είναι πολύ ε, περισσότερο για τους νέους γεωργούς από ότι για το μέσο όρο. Αλλά είπατε ότι υπάρχουν και εμπόδια για την πρόσβαση σε ε, ενισχύσεις και ότι υπάρχουν και έξοδα συμβολογραφικά, Αλλά παρακαλώ προσέξτε κάτι και το είπατε ότι είσαστε και οικονομολόγος ε, ε φιλελεύθερη ρεύματο. Εντάξει, δεν σα κατηγορώ. Αλλά τι γίνεται εδώ. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το χειρότερο ότι μακροπρόθεσμα δεν ξέρουν τι γίνεται γιατί για 20-30 χρόνια πρέπει να επενδύσουν να δουν και τα αποτελέσματα και δεν αναφέρεται την χρόνια ε, αυξανόμενη αστάθεια. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν, χειροτερεύουν, ε, ε γνωρίζοντα και τους γεωργούς στην περιοχή μου και πολλές φορές όταν πηγαίνω εκεί αυτά μου λένε ότι είναι το υπεριθμό ένα πρόβλημα, ότι είναι η σημερινή πραγματικότητα ίδια με την αυριανή. Άρα λοιπόν αλλάζουν πολλά πράγματα στη γεωργία, εντάξει, ανάλογα με την ε, εποχή, το χρόνο, αλλάζει και η σοδιά, αλλάζουν οι τιμές, είναι ο οικονομικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν βλέπουμε όμως διαφορές, δύο παραδείγματα, η αγορά γάλακτος, ε, το καλοκαίρι του 2007 είχαμε 45-46 λεπτά το λίτρο και το 2009 είμαστε 18 λεπτά στα μισά δηλαδή. Και 130 ο τόνος το σιτάρι, πήγε 130 και μετά υπήρξε και κερδοσκοπία γιατί το καλοκαίρι είχαμε πυρκαγιά στη Ρωσία και πήγε στα 152 ευρώ τον τόνο. Α, λοιπόν, ε, έτσι και έτσι βραχυπρόθεσμα δεν μας έλειπε, δεν μας έλειπε σιτάρι επειδή είχαμε αποθέματα. Αλλά τι γίνεται στις έρευνές σας εσείς ε, ποσοτικές και ποιοτικές ε, αυτά. Είδατε αυτά ότι επειδή δεν ξέρουν τι γίνεται μακροπρόθεσμα, επειδή είναι ασταθείς οι αγορές μακροπρόθεσμα, αυτά αναφέρουν ε, οι άνδρες και γυναίκες αγρότες και αγρότες. Ε, σε αυτό τους ανησυχεί, εντάξει δεν είναι ο ρόλος σας εδώ να δείτε αυτούς τους μηχανισμούς, θα το δούμε αυτό, θα το κάνουμε με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή. Αλλά τι γίνεται, αναφέρθηκε αυτό, είτε διαφέρει η κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη, ορισμένοι άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτές τις αλλαγές της Γεωργίας ε, από άλλους. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τι γίνεται για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε τον Μάρκ Ταραμέλα. Ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου. Εργάζεται, δουλεύει το δικό μου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι νέοι αγρότες, οι νέοι γεωργοί ίσως ε, θα πρέπει να τους αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή όχι μόνο είναι νέοι και δυναμικοί αλλά επειδή μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα, την ε, δροσιά τους, τις ιδέες τους, πολλά και διάφορα καινούρια. Και τώρα πρόσφατα διαβάσαμε μία έκθεση που είχε να κάνει με τις γυναίκες στη Γεωργία, την έκθεση της κυρίας Γέγκε νέοι, οι νέες μπαίνουν σε αυτές τις ειδικέ κατηγορίες και οι νέοι ακριβώς ανησυχούν για τη ζωή τους, για το επίπεδο ζωή τους σε αγροτικές περιοχές. Ε, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να υιοθετήσουμε, τι εργαλεία για να παραμείνουν εκεί, αλλά εάν δεν ε, ασχοληθούμε με την ποιότητα ζωής τους σε αυτές τις αγροτικές περιοχές δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρόκειται για τις υποδομές, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται ήδη και επίσης οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα χρηματοδοτεί προγράμματα για τον εξυγχρονισμό του κόσμου της Γεωργίας στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα και η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει ακριβώς σε κατάλληλο επίπεδο να χρηματοδοτείται ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αγροτικές μας περιοχές και έτσι να έχουμε και σαν στόχο ε, τους νέους γεωργούς και για το μέλλον λοιπόν της ΚΑΠ χρειάζεται να διατηρήσουμε τις, ε, τους το χαρακτήρα των ενισχύσεων στους νέους. Και οι πρωτοβουλίες αυτές ε, έχουν στεφθεί με επιτυχία γιατί 3.000 νέοι από το 2008 στη Ρουμανία μέχρι σήμερα ε, ευεργετήθηκαν παρόμοιο πρόγραμμα βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε την γραφειοκρατία και η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλα με ένα σύστημα που να ισχύει σε μόνιμο χαρακτήρα και όχι στιγμία εδώ και εκεί. Και θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς την εγκατάσταση νέων γεωργών αλλά και νέων που ζουν σε αστικές περιοχές και που μπορούν να, με, να πάνε σε αγροτικές περιοχές και να ξεκινήσουν μια αγροτική σταδιοδρομία, την αποκαλέσουμε έτσι. Εδώ λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν, ελπίζουμε ότι έτσι θα βοηθηθούν οι γεωργοί και να μπορέσουν να πάρουν τη σκητάλη και να ασχοληθούν με τη γη επιτέλους. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικουλέσκου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Dorfman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό το workshop σήμερα είναι πολύ σημαντικό γιατί πράγματι αν δούμε την κατάσταση στην Ευρώπη πολλά κράτη-μέλη δεν θα έχουν νέους παραγωγούς στο μέλλον δεν είναι εξασφαλισμένη η επιβίωση της ΚΑΠ. Τι νόημα έχει η ΚΑΠ όταν δεν θα υπάρχουν νέοι γεωργοί. Γι' αυτό το θέμα του σημερινού εργαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη. Και ήδη ελέγχθη ότι πρόκειται για την ελκυστικότητα αυτού του τομέα. Και όταν λέμε ότι ένα επάγγελμα μία απασχόληση είναι ελκυστικό, μιλάμε για οικονομικά ωφέλη. Και θα πρέπει να το καταστήσουμε χρηματικά, οικονομικά ελκυστικό για να κρατήσουμε τους νέους παραγωγούς. Εγώ προέρχομαι από μία περιφέρεια όπου η διαχείριση της γεωργίας ε, είναι δύσκολη. Όμως δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόβλημα με νέους παραγωγούς διότι έχουμε αρκετούς, έχουμε μια, έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη ποιότητα της ζωής, τις παρεχόμενες βασικές υπηρεσίες, το εισόδημα, τη διασκέδαση, όλα. Ε, για να μπορέσουμε να πείσουμε τους νέους να παραμείνουν στην Ήπεθρο. Η ανάπτυξη της ε, Ήπεθρου γενικά είναι ένα μεγάλο τομέα ε, για να μην φεύγουν οι νέοι όλοι στις πόλεις. Επίσης, μέσω του Εράσμους πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε προγράμματα ανταλλαγής νέων αγροτών, νέων παραγωγών, Επίσης τα πανεπιστήμια και η εκπαίδευση γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να συνεργαστούν διότι σε, πολλές, ε, σε πολλούς τομείς αναπτύσσουν αγροτικές πολιτικές. Επίσης η παραγωγή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να, ε, εκπονήσουν, να, να συνεργαστούν για να εκπονήσουν προγράμματα. Πιστεύω ότι στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής πρέπει να σκεφτούμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα διευκολύνουν την ε, παράδοση, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων παραγωγικών ή την συνέχιση των υπαρχουσών παραγωγικών μονάδων από γενιά σε γενιά. Ε, πολλές φορές οι εκμεταλλεύσεις σταματούν να λειτουργούν διότι η παλιά γενιά, η παλαιότερη γενιά δεν θέλει να τις κληρονομήσει, δεν θέλει να τις δώσει στα χέρια των νέων. Θα πρέπει ίσως λοιπόν να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους παλαιότερους ε, γεωργούς, για τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς να παραδώσουν τα ενία σε νεότερους πρόορη συνταξιοδότηση ενδεχομένω, άλλα οικονομικά κίνητα για να παρατηθούν, να αποσυρθούν από τη δουλειά αυτή, για να καταλάβουν επιτέλους οι πιο μεγάλοι αγρότες ηλικία ότι πρέπει να δώσουν τα ενία στους νεότερους. Ευχαριστούμε. Κανιέται. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ζητήματα συζητήσαμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Παραδείγματο χάρη, αν θα μπορέσει να αναπτυχθεί το ευρωπαϊκό δυναμικό με ποιοτικά μέτρα. Ε, έχουμε τώρα ε, βεβαίως μελετήσει επισταμένο στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Γι' αυτό πρέπει να μελετήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα πώς μέσα στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα μπορούμε να βρούμε μέσα για να ενισχύσουμε τους νέους παραγωγούς. Και δι, στην εκπαίδευση, καταρχάς, στην κατάρτιση, στην ε, δημιουργία της αγροτικής υποδομής, τις κατάλληλες επενδύσεις και άλλα ε, συναφή μέτρα. Ήθελα να ε, θέσω το, το, θέμα της αγοράς γεωργικής γης, της αγοράς της γης από νέους αγρότες. Αυτήν ε, Λετο, Λετωνία οι, οι καταβολές ανά εκτάριο γεωργικής εκμετάλλευσης είναι οι ελάχιστες, είναι μικρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ε, συζητήθηκε το πρόβλημα ε, στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Λετωνίας ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ενοικίασης γεωργικών γεών διότι η ενίσχυση που δίνεται είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και επίσης ότι στη Λετωνία δεν επιτρέπεται η πώληση αγροτικών γεών σε άλλους υπηκόους ή σε άλλων κρατών μελών. Τώρα όμως παρόλο που υπήρχε διάθεση αγοράς από άλλους ε, υπηκόους, η τιμή της αγροτικής γης έχει αυξηθεί τόσο πολύ ώστε πάλι να μην μπορούν να την αγοράσουν. Και από την άλλη πλευρά, οι, οι ντόπιοι παραγωγοί, οι νέοι, δεν μπορούν και αυτοί να αγοράσουν τη γη, διότι δεν έχουν κατάλληλα, την κατάλληλη οικονομική ενίσχυση. Ε, υπάρχει λοιπόν μεγάλο πρόβλημα στην τιμή της αγροτικής γης ε, και στην ε, αγορά για, για ιδιοκτησία. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν που εμποδίζει την ε, ελκυστικότητα ε, αυτής τη απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να τα σκεφτεί αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δει πω μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Οι γεωργοί σε άλλα κράτη-μέλη έχουν μια σημαντική συμβολή στα οικονομικά δεδομένα, στην οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να ενισχύσουμε το εισόδημα των νέων παραγωγών και να δοθούν ειδικέ τιμές στα προϊόντα ε, των νέων παραγωγών. Το πρόβλημα στη Λετωνία είναι έντονο. Πώς μπορούμε να χειριστούμε το δημογραφικό και πώς μπορούμε ε, να προσελκύσουμε περισσότερους νέους στον τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Κανιέτε. Σέβερ τώρα. Είχα την τιμή να υποδεχθώ νέους αγρότες από τη Σλοβενία και μου είπαν ότι συμμερίζονται το ίδιο πρόβλημα όπως και οι συνάδελφοί τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γυναίκες και νέοι είναι οι δύο ευαίσθητες ε, ομάδες, ιδίως στις πιο παραδοσιακούς τομείς ε, της γεωργίας. Ε, όταν μιλάμε για προσέλκυση, όταν μιλάμε για ελκυστικότητα του τομέα, η γεωργία έχει παρόμοια προβλήματα, όπως και άλλα επαγγέλματα παρόλο που είναι αναγκαία στην ευρωπαϊκή οικονομία, δεν έχουν ε, τόσο μεγάλη ελκυστικότητα. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν και πιστεύω ότι ο αγροτικός τομέας δεν θεωρείται πλέον ίσονος ε, σημασίας. Πολλοί άνθρωποι ζουν καλύτερα στην Ήπεθρο, σε αγροτικές περιοχές, από ότι στις πόλεις. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, αν κάποιος μου έλεγε είμαι γεωργός, ε, είμαι γεωργός, τον κοιτούσε έτσι λίγο με καταφρόνηση. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Πάντως, εγώ υποστηρίζω τις ιδέες του Πρόεδρου των νέων ε, γεωργών, ε, των νέων αγροτών και υποστηρίζω επίσης και την ε, δραστηριοποίηση του Εράσμους, του Λεωνάρντο και άλλων παρεμφερών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η νέα ΚΑΠ μας απασχολεί πολλές φορές. Και ναι, οι παραγωγοί μας λένε ότι πρέπει και αυτοί να καλύπτονται. Πρέπει λοιπόν να τους καλύψουμε σε όλες αυτές, να συμπεριλάβουμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ τώρα. Σας Γουτιέρες. Ναι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι και αυτό εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για το μέλλον της γεωργίας και της ΚΑΠ. Ο στόχος της είναι να εγγυηθούμε για την παραγωγή αυτή. Θα πρέπει να δούμε, να βοηθήσουμε εκείνους που θα εγγυηθούν αυτή την επάρκεια στο μέλλον και τη νέα γεωργία, το νέο γεωργό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας απασχολεί ιδιαίτερα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μιλάμε και πάλι για τη γεωργία σαν μια ε, σαν ένα χώρο με τη δημιουργία θέσεων, θέσεων εργασίας όπως και στην και με στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας. Αποτελούν όλα αυτά μια ευκαιρία για τη γενιά μας. Βλέπουμε την κρίση την οικονομική, ότι υπάρχουν και περισσότεροι άνεργοι νέοι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα, κάτι που θα ελξει τους νέους και να αποφύγουμε πια την ανεργία των νέων και όπως τον είπαν και άλλοι και οι πυρογνώμων και ο πρόεδρος του ΕΝ Σέντζα για να δούμε πώς θα εγκατασταθούν αυτοί οι νέοι χρειάζεται να προσέξουμε και την πορεία της γεωργίας, την ανάπτυξή της, όλα αυτά τα γενικά που έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο σημεία της αλλαγές, όπως είπε και ο Ταραμπέλα, ε, Επαρκέ εισόδημα, τη δημόσια υπηρεσία, τι επικοινωνίε, το εισόδημα βέβαια. Όλα αυτά είναι σημαντικό για την εγκατάσταση εκεί των νέων για μια ισχυρή γεωργία, για μια ισχυρή γεωργική πολιτική και μια ικανοποιητική γεωργική ανάπτυξη. Υπάρχουν σημαντικά σημεία, συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται υπέρ των νέων. Εδώ έχουμε ε, το κεφαλαίο κινδύνου, διευκολύσεις στις πιστώσεις, ε, στα δάνεια, Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις πολιτικές που είναι πολύ σημαντικές, μπορούμε εκεί να επηρεάσουμε στο μέλλον της ΚΑΠ. Θα πρέπει να δούμε την στήριξη για την εγκατάσταση και άκουσα ότι το να περάσει κανείς από το δεύτερο πυλώνα στον πρώτο πυλώνα δεν ξέρω αν γίνεται αυτό από τεχνικής πλευράς. Είναι όμως κάτι το πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουν τα πράγματα στο δεύτερο πυλώνα να δούμε τα μέσα αντίπια προοριτικά να είναι δεσμευτικά ή Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ακούσαμε και τα στοιχεία από την εμπειρογνώμονα για τις περισσότερες, για τις μεγάλες χώρες, Γερμανία και Γαλλία, που πάνε περισσότεροι εκεί σε αυτούς τους δύο τομείς κτηνοτροφία, γεωργία και υποστηρίζουν περισσότερο αυτό το μέσο του δεύτερου πυλώνα με 140.000 ευρώ σαν βοήθεια για την εγκατάσταση νέων εκεί απέναντι σε χώρες από την Ανατολική ας πούμε Ευρώπη που δεν αφιερώνουν πολλά χρήματα για να αποτελέσει μια πολιτική με πραγματική βούληση διάθεση για αυτήν την εγκατάσταση. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια αύξηση του ποσού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βοήθεια προς τους νέους ε, αντί για 50-50 να είναι 80-20 και 90-10 ε, από πλευρά των κρατών και για να υποστηρίξουμε τους νέους και στη γεωργία πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, να τους καταρτήσουμε. Αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ενσωματώσει και αυτή την έννοια την διαβίου μάθηση και ε, στην κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και να το έχουμε κάτι το μεμονωμένο αυτό. Αφού όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τους νέους αλλά και όλους τους γεωργούς κατάρτιση και όσον αφορά την ε, γεωργία, αλλά παντού και γύρω, για να περισσότερη αποτελεσματικότητα για καινοτομία, για την εμπορία των προϊόντων και την διαπραγματευτική θέση και την διάρκεια των αγροκτημάτων σε αυτό το τομέα. Εδώ, σε αυτό το δεύτερο, θα, το δεύτερο πυλώνα για την κατάρτιση και διαβίου κατάρτιση θα πρέπει να δούμε και να πω κάτι ακόμα, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΘΕΧΑ, ε, σχετικά με τον ε, κόσμο που αποχωρεί ε, συνταξιδοτούμενος. Εδώ έχω ορισμένε αμφιβολίες. Τι είδα τα τελευταία χρόνια ότι πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξυπηρέτησε η πρόορη συνταξιότηση για την εγκατάσταση νέων. Εδώ λοιπόν δεν ξέρω στον τομέα αυτό, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προσθέσει κάτι και αν θα υπάρξουν νέοι που θα εγκατασταθούν και θα αυτή την ε, αυτή την ε, δραστηριότητα. Πάντως ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο για την ποιότητα της εργασίας τους. Ευχαριστώ Σέρτζιο Λεοπρόεδρος. Ανιώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να πει είναι ότι πάντοτε κάποιος θα εμφανιστεί από το πουθενά να καλλιεργήσει τη γη εφόσον υπάρχει κέρδος. Άρα λοιπόν η κερδοφορία είναι σημαντική. Θέλω να διαχωρίσω την ε, γεωργική παραγωγή σε δύο τομείς. Τις καλλιέργειες και τις εκτροφές. Στο Ενωμένο Βασίλειο καλλιεργήσιμη αξία της γης είναι περίπου 80.000 ευρώ ανά εκτάριο. Δεν μπορεί όμως κανείς να την αγοράσει και να την εκμεταλλευτεί ταυτόχρονα, διότι συνήθως την αγοράζουν για επενδυτικούς λόγους και κρατάνε τη γη. Άρα, το να δώσουμε μεγάλα χρηματικά ποσά σε κάποιον για να αγοράσει γη, πιστεύω είναι άσκοπο. Ο συνήθις τρόπος είναι η κληροδότηση η γη κληρονομιέται. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο πλάγια και όχι κάθετα. Όπως αναπτύσσεται η τεχνολογία, έτσι αναπτύσσεται και η τεχνολογία. Και πολλές φορές οι αγροτικές μονάδες ε, τις διαχειρίζονται 4-5 ε, παραγωγοί μαζί. Κάνουν δηλαδή μία κοινοπραξία, μία εταιρεία. Και διαχειρίζονται από κοινού αυτήν την εκμετάλλευση, μοιράζονται τα μπόνους ε, ε, χωρίς να, ανήκει, να τους ανήκει η γη. Από την άλλη πλευρά τώρα της ε, εκτροφής και της βοσκής. Ένας παραγωγός ο οποίος έχει πρόβατα και βοηθεί προσλαμβάνει προσωπικό. Και λέει κάποιο, ναι, θα έρθω να σε βοηθήσω στην μονάδα εκτροφή, αλλά θέλω και εγώ να έχω μερικά ζώα δικά μου. Άρα, αυτό σημαίνει ότι ο νέο παραγωγό θέλει τη δυνατότητα να έχει ένα μισθό και να δημιουργήσει μια μικρή δική του μονάδα. Η δυσκολία που υπάρχει είναι στη στέγαση, διότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις ε, μονάδες θέλουν να μένουν εκεί πέρα αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει απαραίτητη ε, στέγη, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα σπίτια. Αυτό βεβαίως είναι πρόβλημα της τοπικής αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε στα τοπικά συμβούλια πολλά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προσέλκυση νέων παραγωγών όπου η δημόσια γη μοιραζόταν και δινόταν για μια χρονομερισματική μίσθωση σε νέους αγρότες. Όμως τελικά το πρόγραμμα αυτό ε, δεν είχε επιτυχία διότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά ε, ε, τους δόθηκε ένα μικρό, ε, μικρές εκτάσεις για να τις καλλιεργήσουν ή να τις χρησιμοποιήσουν δεν είχαν κέρδος δεν, ήταν, μπορέσαν, να τις εκμεταλλευτούν και δεν είχαν επαρκή κερδοφορία για να παραμείνουν καλή ιδέα λοιπόν αλλά τα προκτικά αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε λεφτά για την αγορά γης Απ' την άλλη πλευρά μπορούμε να δώσουμε χρήματα αν θέλετε στους εκτροφείς όσα θέλετε χρήματα αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το Μερκοσούρ. Πολλοί θέλουν να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ, οπότε θα τραβήξουμε το χαλί κάτω από τα πόδια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Νιώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, και να συγχαρώ τους νέους ε, παραγωγούς για την ε, δέσμευση που έχουν έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αγροτικής, του αγροτικού τομέα. Έχω και παρατηρήσει και ερωτήσεις. Πιστεύω ότι η προσέγγιση προς ε, την ε, αγροτική εκμετάλλευση έχει αλλάξει. Παλαιότερα ήταν υποβαθμισμένη η γεωργία, ε, αλλά τώρα το επάγγελμα αυτό έχει αναβαθμιστεί. Έχουμε και όλα τα θέματα της ασφάλειας των τροφίμων που έχουν επικεντρώσει την προσοχή στη γεωργία περισσότερο όταν ρωτήσεις ε, μια ομάδα νέων πόσοι από εσά θέλει να είσαστε γεωργοί, πολύ λίγοι θα σηκώσουν τα χέρια τους. Ή αν ρωτήσεις αν θέλουν να γίνουν πολιτικοί στο μέλλον, πάλι λίγα χέρια θα σηκωθούν. Ε, η δυσκολία τώρα της ιδιοκτησίας της γης ε, είναι μεγάλη. Καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε ως νέο, νέο αγρότη. Ε, ε, εντάξει, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ νέα όταν κοιτάω τον καθρέφτη πολύ ευχαριστημένη αλλά ε, <laughs> ευχαριστώ πρόεδρε για το κομπλιμέντο σας απλώς ήθελα να σας τσεκάρω αν με παρακολουθείτε λοιπόν το θέμα των πληρωμών, των πιστώσεων, εάν θα διαθέσουμε ένα μέρος από τις διαθέσιμες πιστώσεις στους νέους αγρότες, πρέπει εκτός από την ηλικία να δούμε και το θέμα της χρονικής διάρκειας. Πότε θα πληρωθούν, για πόσο χρονικό διάστημα και πότε θα σταματήσουν οι πληρωμές όταν δεν θα είναι πια νέοι. Η ιδέα λοιπόν τη δημιουργία ενό αποθέματο, αυτό υπάρχει σε ορισμένα κρατημέλη. Μπορεί να μην είναι επαρκή, αλλά υπάρχει Ω εργαλείο, ω μέσον. Στην Ιρλανδία είχαμε δύο προγράμματα προώρης συνταξιοδότησης και ενίσχυσης νέων παραγωγών και ήταν αποτελεσματικά τα προγράμματα. Όμως το πρόβλημα με το δημόσιο, με τις δημόσιες πληρωμές είναι, και την κρίση είναι τα προγράμματα αυτά έχουν εγκαταλειφθεί και έτσι δεν υπάρχει συνοχή και συνέχεια στις πολιτικές αυτές. Ο κύριος Σάγνιου πιστεύω ότι έσυσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Εάν ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τον αγροτικό τομέα με νέους παραγωγούς πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τα προβλήματα των αγορών, για την αστάθεια στις αγορές, να βρούμε μέτρα ενθάρρυνσης των νέων χρειάζεται να γίνει αυτή η μεταφορά από γενιά σε γενιά. Πρέπει να παραδοθούν ε, μονάδες στα χέρια νέων. Και επίσης να ενισχυθεί η θέση των γυναικών. Ευχαριστώ. Υπέροχο, υπέροχο, Μαρέδ, Ο Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη, εγώ ήμουν στην Επιτροπή από δίπλα ε, μέλος. Εδώ αυτό το θέμα μπορεί να καταλήξει σε αυτόν τον αριθμό 7% κάτω των 35%. Ορισμένοι είμαστε στην Επιτροπή για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές ε, και Είδαμε την επίθεση κατά του προπολογισμού τη Γεωργία. αυτή ο αριθμό των 7% δικαιολογεί ότι η ΚΑΠ ε, δικαιολογείται και παρόλα τις προκλήσεις 2014-2020 ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε την ανανέωση των γενεών εντάξει θέλετε να λέμε για την προμήθεια τροφίμων, για την αυτάρια κλπ. Αν δεν έχουμε κάποιον να δουλέψει για αυτή την ανανέωση δεν θα έχουμε και αποτελέσματα. Απλά και μόνο θα ήθελα ένα ερώτημα να θέσουμε. Στη γεωργική ανάπτυξη, στον προγραμματισμό υπάρχουν πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την εγκατάσταση των νέων εκεί. Και στα εργαλεία αυτά έχουμε τη σελίδα 4041 πάρα πολλά που, δάφια που δείχνουν ότι χρησιμοποιούν αρκετές χώρες αυτά τα εργαλεία. Εντάξει, τι βλέπουμε και μέσω του προπολογισμού και μέσω των αριθμών ότι λίγες ε, χώρες έχουν μια πραγματική πολιτική με βούληση απέναντι σε την εγκατάσταση επιτροπή. Μας ίσως θα πρέπει εκεί να το προσέξει λεπτομερέστερα, να καταλάβουμε το γιατί, να δούμε πώς αυτά τα εργαλεία δείχνονται εδώ αποτεσματικά και εκεί όχι και θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε μια πολιτική με ένα δεσμευτικό μέρος αλλά του δευτέρου πυλώνα πολιτική, γιατί η κοινωνική πολιτική και η φορολογική πολιτική, τα δικαίωμα διοκτησία και οι κληρονομίε κλπ. Όλα αυτά είναι διαφορετικά. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να το βενταχθούν στον πρώτο πυλώνα, ενώ στο δεύτερο πυλώνα μα επιτρέπει να διαθέτουμε εργαλεία που είναι τα καταλληλότερα σύμφωνα και με τα εθνικά διαφορετικά δίκαια. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Λέω Πρόεδρο. Σκότα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μ, άκουσα αρκετές παρεμβάσεις ε, από αρκετούς συναδέλφους. Ε, εντάξει, συμφωνώ, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά. Να πω όμως, να επιμείνω ότι για την κατάρτιση ήδη από την αρχή από το σχολείο, τη βασική εκπαίδευση, είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει να το ευαισθητοποιήσουμε, να βεθούν αυτά τα παιδιά ότι η γεωργία είναι ένα τομέα ενδιαφέρον ε, το γενός και αυτό το βγαίνουν από εκεί μπορεί να είναι κάτι το σημαντικό. Αυτό μερικές φορές και στην Ιταλία, τη δικιά μου τη χώρα, το λησμονούμε. Και βέβαια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι αρκετοί νέοι και θα πρέπει να δείξουμε αυτή την ευαισθησία και όσοι δεν πιστεύουν. Ακούσαμε την εισηγήτρια που μίλησε για ορισμένα προβλήματα, προβλήματα των νέων που δεν θέλουν να εγκατασταθούν εκεί για πολλούς λόγους. αλλά λοιπόν, είναι ευαίσθητοι και μπορεί να δημιουργηθεί και μια ευαισθησία ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την εγκατάλειψη διαφόρων περιοχών, δύσκολων ίσως, και ότι δεν χρησιμοποιούνται πια οι περιοχές αυτές που δημιούργησαν μια σημαντική γεωργία στο παρελθόν, όχι τώρα όμως δυστυχώς, και που οφείλεται και στο ότι ορισμένοι φορείς και εθνικοί φορείς με διάφορες ρυθμίσεις και νόμους και που τελέχουν τα πράγματα. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε κάτι, να προστατεύσουμε και την ύπεθρο και όχι να χρησιμοποιήσουμε τη γη έτσι κερδοσκοπώντας γιατί βλέπουμε παντού ότι έχουμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που δεν έχουν τίποτα, καμιά δουλειά εκεί πέρα. Ε, παντού έχουμε ε, αιωλικής παραγωγής ε, εγκαταστάσεις και όλα αυτά για μια σωστή, καλή παραγωγή, καλή ποιότητα, αλλά για και εκείνους που μετά θα πρέπει να διαθέτουν άθικτες αυτές τις περιοχές για να τις εκμεταλλευτούν. Εδώ στην περίπτωση αυτή επειδή αλλάζει, μεταβάλλεται η τεχνολογία, σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, μια, κάποια ογκομετρία σε αστικό επίπεδο παντού και θα πρέπει ο γενής τομέας ε, θα πρέπει να συνδυαστεί με ορισμένες παρεμβάσεις ε, που έχουν να κάνουν με την ίδια τη δουλειά, την εργασία και όχι να λέμε ότι είμαστε ανώτεροι και ρυθμίζουμε τις καταστάσεις χωρίς να καταλαβαίνουμε αυτό που ζητείτε όγκομετρικά και να βλέπουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που θα πρέπει να τα βολεύουν όπως όπως και να ε, παρανομούν και όσον αφορά τα κτίρια τους. Ναι, κλείνω η συζήτηση. Έχεις το λόγο. Ε. Ε, κυρία καθηγήτρια, ασχοληθήκατε με το θέμα της μόρφωσης των νέων αγροτών. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω η μόρφωση είναι καλύτερη. Είδατε τα αποτελέσματά τους ή μήπως ε, ξέρετε αν οι νέοι αγρότες έχουν καλύτερα, καλύτερες επιδόσεις. Επίσης, το, μέλ, το μέγεθος των αγροτικών γενιών. Είναι πιο πολύ άρδινες από τις αστικές οικογένειες. Και επίσης, μήπως βλέπετε κάποιες τάσεις οργάνωσης των νέων αγροτών μεταξύ τους, γιατί μία ε, από τις πληγές της ε, ε, γεωργικής ζωής είναι η έλλειψη οργανώσεων. Απλώς οι νέοι παραλαμβάνουν τη γη των γονιών τους. Μήπως υπάρχουν περιπτώσεις που η επιλογή του επαγγέλματος γίνεται εντελώς ανεξάρτητα. Δηλαδή κάποιος εκτός της υπαίθρου, κάποιος κάτοικος πόλης έχει κάνει μια πραγματική επιλογή επαγγέλματος, έχει επιλέξει να γίνει αγρότης ή είναι αυτό σπάνιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεκερεύσκη. Το λόγο έχει τώρα η καθηγήτρια Ζαβαγόσκα και μετά για λίγα λεπτά και ο πρόεδρος του ΣΕΖΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σικέρσκι ιδιαίτερα για την ερώτησή του. Γνωρίζετε πολύ καλά, πιστεύω, την κατάσταση των νέων αγροτών στην Πολωνία από άποψη μόρφωσης και κυρίως ε, όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Είχαμε στοιχεία για όλους τους ε, αγρότες. Δεν χρησιμοποίησα δεδομένα από ερωτηματολόγιο ή άλλα στατιστικά δεδομένα. Έχω όμως μια, έναν απλό πίνακα μέσα στην έκθεσή μου που αφορά τη σύγκριση του αριθμού των αγροτών με μόρφωση ανωτά του επίπεδου, κυρίως σε θέματα γεωργικής παραγωγής. Το έβαλα για διάφορους λόγους. Καταρχήν επειδή ένα από τα βασικά εμπόδια της παραλαβής από τους νέους αγρότες ε, του κλήρου των γονιών είναι, η έλλειψη, είναι το θέμα της ανώτατης παιδείας. Δηλαδή, πολλοί που θα μπορούσαν να κληρονομήσουν ή να αναλάβουν από τους γονείς τους, ε, να παραλάβουν τη γη, δεν έχουν τέτοιου είδους μόρφωση αγροτικής οικονομίας. Συνέταξα λοιπόν ερωτηματολόγια και τα έδωσα σε 200 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας. Κάναμε και μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας και πριν έρθω εδώ συζήτησα σε με τέσσερις ομάδες και ρώτησα αυτούς που προέρχονται από την Ήπεθρο και οι οποίοι θα μπορούσαν να παραλάβουν ε, τους, από τους γονείς ε, τους είπα και μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το εμπόδιο. Γιατί λοιπόν δεν επιλέξατε ένα πτυχίο που θα σας οδηγούσε σε τέτοιου είδους μόρφωση. Α, είπαν ότι θέλαν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βρουν μια καλή δουλειά. Γιατί αν σπουδάσω γεωπόνος ή αγροτική οικονομία, μόνο σε αυτόν τον κλάδο θα μπορώ να δουλέψω. Ενώ αν μορφωθώ και αποκτήσω μια άλλη παιδεία, ένα άλλο πτυχίο, ίσως θα είναι πιο εύκολο για μένα να βρω μια θέση αλλού. Αυτή ήταν η απλό απάντηση στην ερώτησή μου. Τώρα, όταν τους, όσον αφορά την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ε, εκμεταλλεύσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αυτό είναι κάτι που δεν μελέτησα, πιστεύω όμως ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε. Το αν και κατά πόσον υπάρχει τάση οργάνωσης ε, των νεαρών αγροτών μεταξύ τους, ούτε ε, τέτοιες τάσεις υπάρχουν φοβάμαι. Στην Πολωνία η εμπειρία μας ε, από τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες καλλιεργητών είναι κακή. Βεβαίως οι νέοι δυναμικοί αγρότες ε, συστήνουν τέτοιου είδους ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Μπορούν να οργανωθούν. Όμως, αν σας ε, πω την κατάσταση στο δικό μου χωριό, και αν ρωτήσετε εκεί τους αγρότες αν θέλουν να συνεταιριστούν θα σας απαντήσουν σαφώς όχι γιατί στις περισσότερες περιοχές η δομή της παραγωγής ε, ε, είναι τόσο διαφοροποιημένη ώστε υπάρχουν αγρότες που παράγουν τα πάντα, άλλοι που δεν παράγουν τίποτα και απλώς παραλαμβάνουν τις ενισχύσεις. Μια δημιουργία λοιπόν ομάδας που εξειδικεύεται σε ένα προϊόν θα είναι πολύ δύσκολο. Ε, συνεταιρίζονται λοιπόν μόνο μόνον όχι ως παραγωγή αλλά ως νέοι αγρότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας. Αυτό το διαπιστώνουν και οι κοινωνιολόγοι. Η, η πολιτική κινητοποίηση των νέων λοιπόν είναι δυστυχώς πολύ δύσκολη. Ίσως αν υπάρξουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα Η δράση λοιπόν για κινητοποίηση, δραστηριοποίηση, στήριξη των νέων ηγετών, ίσως κάτι θα πέδιδε. Όσον αφορά τώρα την το την μετακίνηση από τις αστικές στις αγροτικές περιοχές, ήδη απίτησα. Δεν μπορώ τα αποτελέσματα που έχω να τα γενικεύσω. Θεωρώ όμως ότι οι κάτοικοι των πόλεων είτε ε, ε, ε, ε, σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο και λένε μάλιστα γιατί να πάμε στις αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν τα παιδιά των αγροτών που πολύ εύκολα μπορούν να μείνουν εκεί. Υπάρχει λοιπόν η πεποίθηση ότι εν... ενώ με μεταναστεύουν ε, τα παιδιά των αγροτών προς τις πόλεις. Η άλλη πλευρά, οι νέοι της πόλης δεν το θεωρούν, θεωρούν την αντίστροφη κίνηση δυνατότητα. οι περισσότερες απαντήσεις που μου έδωσαν αφορούν το επίπεδο ζωής. Ίσως είναι πολύ νέα αυτά τα παιδιά, κάποιοι είναι ακόμα κάποιοι εργάζονται ε, και παράλληλα σπουδάζουν και τους ενδιαφέρουν περισσότερο άλλα, άλλα πράγματα, η κοινωνική ζωή, η ψυχαγωγία, ποιότητα ζωής κλπ. και από τα οποία δεν θέλουν να παραιτηθούν. Πέραν αυτό, νομίζω ότι και τα χρήματα αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξουν. Αυτό το οποίο επανειλημμένως αναφέρθηκε είναι η δουλειά σε επίπεδο βάσης από νεαρή ηλικία. Πρέπει κανείς να ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια του σχολείου να ε, διαφημίζει, να διαδίδει αυτή την ιδέα ε, στους νέους μαθητές. Γιατί πολλοί νέοι δεν θεωρούν μόνο ότι το να είναι κανείς αγρότης πάει το ότι είναι ένας αμόρφωτος χωριάτης, ε, ε, αλλά και άλλα τέτοια σχετικά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τα νέα παιδιά, αλλά και τους τοπικούς ηγέτες κλπ. κλπ. Απαντώ στην ερώτηση και σχεδόν τελείωσα. Μάλλον τελείωσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Νέων Γεωργών έχει το λόγο για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ ε, και μπορώ να παρακολουθήσω τα σχόλια και τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών που αντιμετωπίζουν την κατάσταση την οποία θεωρούν ανησυχητική ή μια κατάσταση που εν πάση περιπτώσει πρέπει να την ε, φροντίσουν. Πραγματικά αυτό ενισχύει την άποψή μας ότι πραγματικά είστε εταίρος μας στην προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος των νέων αγορωτών στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Ε, ο κύριος Καραμπέλα ε, ρώτησε κάτι για την ε, τις είναι κάτι που και εμείς ε, το μελετάμε και η κυρία ε, Μαγκίνης το ρώτησε αυτό ναι ρίτε. Ε, πρέπει να το κοιτάξουμε σήμερα η κατάσταση των νέων αγροτών είναι συγκεκριμένη αλλά στις συνεδριάσεις και στα σεμινάρια που οργανώνουμε εξετάζουμε και την κινητικότητα της αγοράς και αυτό είναι ένα από τα θέματά μας ενδεχομένως την επόμενη φορά να σας παρουσιάσουμε σκέψη για αυτό το θέμα. Είναι πολύ ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι πολλοί από εσά ε, υπογραμμίσατε τη σημασία της κατάρτισης, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα επίπεδα της ε, εκπαίδευσης, αλλά και η οποία να συνεχίζεται μέχρι και τη φάση που ξεκινά κανείς ε, την επιχείρησή του. Γι' αυτό προτείνουμε αυτά τα κουπόνια γνώσης που θα διανέμονται στους νέους αγρότες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον δε και το πρόγραμμα Εράσμους που θα απευθύνεται συγκεκριμένα σε νέους αγρότες που μπορούν να ταξιδεύουν για να μάθουν. Αυτό θα ενισχύσει τις γνώσεις τους για την ΚΑΠ αλλά και τις γνώσεις τους για τις διαφορετικές μορφές, την πολυμορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ο κύριος Νικολέσκου ανέφερε το γεγονός ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους ενεργούς αγρότες. Και εμείς το υπογραμμίσαμε αυτό. Η ελκυστικότητα της γεωργίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση ή αναφέρθηκε και από κάποιους από εσά. Σας διαβεβαιώνω ότι τα μέλη των οργανώσεων που εκπροσωπούμε σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ ικανοποιημένοι με το επάγγελμά τους, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πολλοί άλλοι νέοι που θα μπορούσαν να μάθουν την ομορφιά της δουλειάς μας. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε να ε, διαδώσουμε. Και εδώ πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα. Η ανακοίνωση αυτή για την Γεωργία και την ΚΑΠ και το για την Γεωργία είναι κάτι που μπορεί να γίνει, ε, να, να ξεκινήσει στο πλαίσιο μιας εκστρατείας στο μέλλον. Ο κ. Καρνιέτε είπε κάτι για τον πρώτο πυλώνα. Και ε, κάποιοι το αμφισβήτησαν. Και επίσης η ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες αφορούσε το συγκεκριμένο αυτό εργαλείο. Ε, μελετάμε τώρα τις δυνατότητες που υπάρχουν, αν μπορεί αυτό να εισαχθεί και αργότερα μπορούμε να σας δώσουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό των ετών, το ποσό της ε, ενίσχυσης και πολλά άλλα. Νομίζω ότι δεν έχω τίποτα άλλο να απαντήσω. Ευχαριστώ όλους όσοι μου έκαναν, όσοι μου ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά λέει ο Πρόεδρος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, και βέβαια και τους δύο συγκητές μας θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε. Το τέσσερα σημείο είναι ο προπολογισμός του 2011. Μετά από την επιτυχία των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό του 2011 θα πρέπει τώρα να δούμε τις ενδεχόμενες συνέπειες για το γεωργικό προϋπολογισμό και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που ίσως δημιουργηθούν εκεί προβλήματα εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία στο άμεσο μέλλον. Παρακαλούμε την κυρία Μαγκίνες να μας κάνει ένα κάποιο σχόλιο για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και στη συνέχεια να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναλύσει όσο γίνεται καλύτερα το επόμενο σχέδιο με τις προτάσεις για τα θέματα της γεωργίας μετά, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το τελευταίο σας σχόλιο για την ανάλυση που έκανε η Κομισιόν του Σχεδίου Προϋπολογισμού είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να παραμείνουν στην αίθουσα. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις επί του αγρογεωργικού ε, ε, προϋπολογισμού αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θέλω λοιπόν να σας το υπογραμμίσω και ως εισηγήτρια θέλω να ζητήσω την υποστήριξή σας. Έχω παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία και άκουσα και μίλησα ε, σε διάφορους χώρους για να επισημάνω στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν τις σοβαρές επιπτώσεις στη Γεωργία. Χρειαζόμαστε όλοι σας την υποστήριξη σε αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζετε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ε, δεν πήγε καλά για να μην πω τίποτα χειρότερο. Υπάρχουν σημαντικά ε, νούμερα που για το Κοινοβούλιο και τώρα ξεκίνησε ένας, ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο συμφώνησε με το αίτημα του Συμβουλίου η αύξηση να περιοριστεί στο σχεδόν 3%. Αρχικά είχαμε ζητήσει περισσότερο. Αρχικά ε, μάλλον ε, ουσιαστικά τώρα η απέτηση είναι να μειωθεί, έτσι είχε ζητήσει η Κομισιόν, να μειωθεί ο προπολογισμό κατά τέσσερα δις και είχε προταθεί να γίνει μια γενική περικοπή κατά ένα τρίτο στο δεύτερο τίτλο, στον τίτλο 2 αυτό μας ενδιαφέρει εδώ και όπως είπα αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις κυρίως στις πολιτικές υπέρ της υπαίθρου. Θα ήθελα η Κομισιόν να επισημάνει επακριβώς ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις. Τα καλά νέα δεν είναι πολύ σημαντικά αλλά πρέπει να σας τα πούμε, να σας πούμε και τα θετικά. Το, σχέδιο, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού μας παραχωρεί μια αύξηση 10 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα ε, ε, γάλακτο στα σχολεία. Επίσης ένα ποσό για την ε, ε, κρίζωση των ασθενειών, όχι αυτό που είχαμε ζητήσει και επίσης ε, είχαμε κάποια ωφέλη για τα προγράμματα Life Plus. Επίσης υπάρχει το θέμα της εκαθάρισης των λογαριασμών, το οποίο παραμένει όχι όσο μας απασχολούσε, αλλά είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων. Εξακολουθεί να παραμένει αυτό το ζήτημα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και ελπίζω να με καταλάβετε. Όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς για τον προπολογισμό, τόσο λιγότερο θέλει κανείς να υποστηρίξει τον τρόπο λειτουργία του. Ε, τόσο, μπορεί, τόσο λιγότερα καταλαβαίνει κανείς τον τρόπο λειτουργία του. Και γι' αυτό από πλευρά κομισιών υπάρχει, πρέπει να πει στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας πόσο θα επηρεάσει αυτός ο προϋπολογισμός ε, πραγματικά τα κράτη-μέλη, τους αγρότες και τις αγροτικές ε, περιοχές. Δεν θα επηρεάσει εξ όσων γνωρίζω τις, ε, ε, την ενιαία ενίσχυση, αλλά πρέπει να δούμε τι δεσμεύσεις θα αναλυφθούν. Τα είπα αυτά στους συναδέλφους γύρω από το τραπέζι του προπολογισμού, του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κατανόησαν. Αλλά μου είπαν και πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό η Κομισιόν, ότι πολλά κράτη δεν χρησιμοποιούν τον ε, προπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης. Επειδή ο λόγος όμως που έχει γίνει στόχος να περικοπείς αυτός ο προϋπολογισμός είναι επειδή είναι ο, μόνο, είναι επειδή ο είναι ο μόνος προϋπολογισμός που μπορεί από τεχνική άποψη να γίνει αυτός ο προϋπολογισμός. Δεν είναι καλά τα ενόψη των Χριστουγέννων, αλλά πρέπει να τα ξέρετε. Ε, πολεμήσαμε σκληρά και εγώ και ο κύριος Λεβία. Όπως σας είπα, είχαμε μια στήριξη, ε, λόγω, ε, υπάρχουν όμως ελλείψεις κονδυλίων και εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα και οπωσδήποτε θα ήθελα η Κομισιόν να είναι απολύτως σαφής επ' αυτού, κυρίως όσον αφορά τη γραμμή για τον καθάριστο των λογαριασμών. Τα έσοδα που ανέβηκαν στα 540 εκατομμύρια. Και πώς έγινε αυτό. Διότι όλα αυτά τα μελέτησα και δεν τα βρίσκω απολύτως ξεκάθαρα. Δεν, βρίσκω, δεν μπορώ με να καταλάβω πώς καταλήξαμε σε αυτά τα νούμερα. Ελπίζω η Κομισιόν θα μπορέσει να μας το πει γιατί έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Επίσης κατάλαβα ότι υπάρχει η πολιτική θέληση να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα ΙΤΑ. Ε, αλλά πρέπει να μας πει η Κομισιόν πώς θα το κάνει. Ε, αυτό είναι μόνιμη ανησυχία της Επιτροπής γιατί ο, ο προϋπολογισμός ε, της Γεωργίας φοβούμαστε επειδή είναι πολύ εμφανής να γίνει ε, πηγή εσόδων για άλλους προϋπολογισμούς ή άλλες γραμμές και αυτό δεν μας φοβίζει μόνο για του χρόνου. Όταν βλέπουμε τα σχέδια για το δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 Λοιπόν, πιστεύω ότι θα, θα σταματήσω εδώ. Θα ζητήσω όπως και εσείς ζητήσατε να ξεκαθαρίσει η Κομισιόν το, κάποια από τα θέματα που έθεσα. Μοιάζει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο κλπ. έχουν την προθυμία ή την επιθυμία να συμφωνήσουν με τον προβολογισμό πριν το τέλος του χρόνου και εν κατακλείδη θέλω να προσθέσω ότι αποτυχία συμφωνίας θα μας βάλει στη διαδικασία των 12 ε, τιμωρίων 12η τιμωρία και αυτό θα επηρεάσει ας πούμε τις προκαταβολές εκεί που έχουν γίνει προκαταβολές θα υπάρχει πρόβλημα Ιανουάριο, Φεβρουάριο κλπ. Και πρέπει λόγω αυτού να επιτευχθούν συμφωνίες. Είναι πολύ ζωφερά ε, τα μηνύματα ε, από την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε. Να τονίσω και εγώ κάτι, παρακαλώ συνάδελφοι, προσέξτε. Το θέμα αυτό που μας είπε η κυρία Μαγκίνες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα ακούσουμε έναν συνάδελφο Λαβία και μετά τον διευθυντή κύριο Λόγκο και μετά επειδή όλα αυτά επηρεάζουν τα πράγματα βράχει πρόθεσμα όπως μας είπε η κύριε Μαγκίνες για την ε, πληρωμές ε, των πληρωμών. Επειδή όμως ε, υπάρχει και ένα πλαίσιο μετά μακροπρόθεσμο για τις δημοσιονομικέ προοπτικές και τον Επίτροπο Σόλος όταν τον ακούσαμε σε συνέντευξη τύπου μαζί με όλου, τους συντονιστές των ομάδων ε, τονίσαμε ότι η Επιτροπή αυτή, εάν δεν είναι σίγουρη για τον προπολογισμό, δεν θα υιοθετήσει για την ΚΑΠ κανένα νομοθετικό κείμενο. Αναλάβαμε έτσι ιδιαίτερη ευθύνη. Θα πρέπει όμως πάνω σε αυτό το θέμα, πώς να σου το πω, να έχουμε σταθερή, ομοιόμορφη θέση όσον αφορά τη στρατηγική μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ντεγκίνες, τον Δόκτωρ Λάρια και μετά Λόγκο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ μόνο δύο πληροφορίες σε όσα πολύ σωστά είπε η συνάδελφος Μαγκίνες. Πρώτο σημείο. Στη συνάντηση αυτή για τον προβλησμό του 2011 το Συμβούλιο σε σχέση και με την κρίση η οποία χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη ζήτησε το πάγωμα των πληρωμών ε, σε ένα κατόφλι σε σχέση με τον προβλησμό του 2010 των 2,91% αλλά ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφερε τη δυνατότητα να αυξήσει τις υποχρεώσεις ε, όχι σαν πληρωμές επαναλαμβάνω σαν υποχρεώσεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ από τεχνικής πλευράς στήλη 2 κάθε σημείο έχει το ίδιο επίπεδο και πληρωμών και υποχρεώσεων άρα λοιπόν ανάμεσα στα δύο υπάρχει ένα τεχνικό εμπόδιο μια μείωση των πληρωμών ε, έφερε και μείωση των υποχρεώσεων και μόνο για ορισμένα σημεία μπορέσαμε να αυξήσουμε τις υποχρεώσεις εκεί που μπορούσαμε και είχαμε δύο άλλα διαφορετικά θέματα στοιχεία σε αυτό. Δεύτερο τώρα σημείο και με ορισμένε δηλώσεις για την Επιτροπή να ζητήσω ακριβώς για το δρόμο που διανύουμε, που προχωράμε για να προχωρήσουμε στον προϋπολογισμό με μια πορεία ε, fast track έτσι επί που έχει επιταχυνθεί, που να, έχει, που να επιταχυνθεί μέχρι το τέλο τη χρονιάς. Αύριο και μεθαύριο στην Επιτροπή προπολογισμού, θα εξετάσουμε την πρόταση προπολογισμού για το 2011 που μόλις υπέβαλε η Επιτροπή. Ουσιαστικά συμφωνούμε όσον αφορά τους αριθμούς, αλλά ορισμένε πολιτικές προτεραιότητες όπως μια κάποια ευκαμψία ας πούμε ε, απαιτείται ένα κάποιο χτένισμα ακόμα των θέσεων και των μεν και των δε και μια αποδοχή από πλευράς του Συμβουλίου των ε, προτεραιοτήτων ε, που έθεσε το Κοινοβούλιο. Στους αριθμούς όμως βλέπω μια περικοπή πει η πιο συγκεκριμένη στη στήλη 2, στη δεύτερη πρόταση προπολογισμού από πλευρά τη Επιτροπή, έχει να κάνει με την γεωργική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή τι γίνεται μετά από την περικοπή αυτή, τι θα γίνει με τις πληρωμές για την γεωργική ανάπτυξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Τζοβάνι. Ο Διευθυντής Λόγκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρέμβω εδώ σε αυτή τη συζήτηση και μου επιτρέπετε να συμμεριστώ μαζί σας την τεράστια αυτή ανησυχία λόγω της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2011. Ναι, το σκηνικό αυτό είναι ιδιαίτερα αβέβαιο και ίσως ε, δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα ήδη τα είπαμε ποια θα μπορούσε να είναι και ειδικότερα προβλήματα που θα εμφανιστούν ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του 2011. Θα επανέλθω με περισσότερη ακρίβεια στην επιτυχία αυτή. Θα ήθελα όμως ε, ταυτόχρονα να τονίσω το θετικό της παρουσίασης ενός νέου σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011. Αυτό έγινε τις 26 Νοεμβρίου και όπως είπε ο κύριος Λεβία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονες δραστηριότητες, ε, το αναλύει κανείς και ελπίζουμε να ξεπαγώσει η κατάσταση και μάλιστα όσο γίνεται πιο σύντομα. Πριν το τέλος της χρονιάς δε ελπίζουμε να διαθέτουμε ένα προβλήσμα που να έχει εγκριθεί. Για να κάνουμε μια ανάλυση της όλης εικόνας. Ε, πώς θα μπορούσα να μη όλα αυτά να μην ε, εγκριθεί ο προπολογισμό. Αυτό με τα προσωρινά δωδεκατημόρια, με ένα περιορισμό του προπολογισμού που θα μπορούσε να θίξει ιδιαίτερα την εκτέλεση της πολιτικής, την άξιση πολιτικής και ιδιαίτερα της γεωργικής πολιτικής όσον αφορά μέτρα. Ευτυχώς, όσον αφορά τα μέτρα της αγοράς, δεν προβλέπεται η εφαρμογή των προσωρινών δωδεκατομμυρίων να οδηγήσει σε ιδιαίτερα προβλήματα γιατί όλα αυτά διανέμονται, κατανέμονται μάλλον ε, κατά τη διάρκεια του χρόνου με αρκετά ομοιόμορφο χαρακτήρα. Από την άλλη μεριά όμως ε, για τις ε, Άμεσε ενισχύσει. Υπάρχει ήδη μια, μια ιδιαίτερη συγκέντρωση από την 1η ε, Ιανουαρίου για τις, για επιστροφές στα κρατημέλη, για τις δαπάνες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για φέτος 11 ε, κρατημέλη τους είχε δοθεί το πράσινο φως να δώσουν ήδη προκαταβολές μέχρι και το 50% της συνολικής ενίσχυσης. Ήδη τον Ιανουάριο, τις πρώτες πρώτες μέρες του Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έλλειψης πόρων για να επιστρέψουμε στα κράτη-μέλη που ακόμα περισσότερο θα χειροτερέψει η κατάσταση και θα ισχύσει για όλα τα 27 κράτη-μέλη τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου. Για να σας δώσουμε κάπως την εικόνα, τη διάσταση και τους σημαντικούς αριθμούς 6,6 δισεκατομμύρια ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος. Βλέπουμε ότι θα έχουμε 31 δισεκατομμύρια ευρώ ποσά. Καταλαβαίνετε πόσο άσκημη είναι η κατάσταση. δίνει και για μας απέναντι στα κράτη-μέλη αλλά και για τα ταμεία των κρατών μελών που σε αυτά τα γενικά πλαίσια κρίσης και έλλειψης πόρων ίσως αντιμετωπίσουν τρομερές δυσκολίες. Για τη γεωργική ανάπτυξη, το πρόβλημα αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να εμφανιστεί τουλάχιστον μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 11. Ε, αργότερα η κατάσταση ε, είναι κάπως ασαφής και αβέβαιη. Και ακριβώς να υπενθυμίσω για να κλείσω το πρώτο μέρος αυτό της παρέμβασής μου ότι ιδιαίτερα ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί από τη στιγμή που θα δείξουμε ότι μαζί κατέχει η αίσθημα υπευθυνότητα, όπω κάνουμε εδώ στα πλαίσια τη νέα συζήτηση για το νέο πρόγραμμα προπολογισμού και ελπίζουμε όλα αυτά να μην ζημιώσουν του γεωργού, οι οποίοι οι γεωργοί επιτακτικά χρειάζονται αυτές τις πληρωμές. Αλλά ούτε και να ζημιώσει τα κράτη-μέλη που ίσως αντιμετωπίσουν δυνα προβλήματα πληρωμών στα ταμεία τους. Αυτά στις γενικές γραμμές της νέας πρότασης του προπολογισμού. Αυτά ήθελα λοιπόν να πω. Και ολοκληρώνοντας την εισαγωγή μου να σας πω ότι ναι αυτή η πρόταση του προπολογισμού όλα αυτά ε, περνάνε στον διορθωτικό στο διορθωτικό που είχαμε κάνει στο πρώτο προσχέδιο του προπολογισμού του 2011 και διάφορα στοιχεία συμβαστικά, προτάσεις συμβαστικές, οι οποίες είχαν άλλωστε προκύψει ε, στα πλαίσια της συνδιαλλαγής. Σχετικά με την αρχική πρόταση, μια από τις κύριες διαφορές είναι κατά 200 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση, όπως έχουν εκτιμηθεί στα πλαίσια της καθάρισης λογαριασμών και της επιβεβαίωσης αυτών και είναι μια αρνητική δαπάνη που σαν συνέπεια θα έχει μια μείωση ενός αντίστοιχου ποσού όσον αφορά τις πιστώσεις η πρόταση της αύξησης των αρνητικών δαπανών για τη γραμμή αυτή προορισμού είχε προταθεί από το Συμβουλίο στην πρώτη φάση εξέτασης της πρότασης της Επιτροπής. Τώρα για να σεβαστούμε και το ανώτατο ποσοστό κατόφλι της αύξησης δαπανών για τον, σε σχέση με τον του 2010, Δυστυχώς ε, υποχρεωθήκαμε σε μια άλλη οδυνηρή περικοπή που δημιουργεί προβλήματα σε αυτά που είχαμε προβλέψει που για την ανάπτυξη της υπαίθρου 214 εκατομμύρια ευρώ όπως το είχαμε άλλωστε αναγγείλει και οι κύριες Μεντίνες και εμείς ε, τι ελπίζουμε, ότι θα εγκριθεί και η πρόταση δήλωσης που ε, προωθήσαμε για να συνοδεύσει αυτή την περικοπή και που οι δύο πλευρές, οι δύο αρχές επί του προπολογισμού, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, να υποχρεωθούν ενδεχόμενα να δουν τις δυνατότητες της ανάπτυξης υπαίθρου ε, όπως πρέπει σε περίπτωση που απαιτηθεί κάτι παρόμοιο. Εδώ, σε αυτά θα ήθελα να περιοριστώ, σε αυτά τα γενικά και η κυρία Μπόρχμαν θα μπορούσε να σας δώσει ορισμένες συγκεκριμένες να κάνει σήμερα για σε συγκεκριμένους αριθμούς. Εντάξει, σύντομα, σύντομα, μετά τη δική μου την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι, νομίζω ότι τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά <clears throat> τα, ε, ε, το, τις, ε, τα έσοδα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι όσο περισσότερο γνωρίζουμε για τον προπολογισμό τόσο πιο ξεκάθαρες είναι οι απόψεις μας, κυρία Μαγκίνες, αλλά έτσι είναι η ζωή. Όσον αφορά τώρα τα έσοδα, έχετε 550 εκατομμύρια carry-over από πέρσι που θα μεταφερθούν στον προπολογισμό του χρόνου, συν 10 εκατομμύρια τα οποία προβλέπονται από την τροποποιητική επιστολή της Κομισιόν. Τα υπόλοιπα 360 εκατομμύρια, 320 εκατομμύρια προέρχονται από την Κομισιόν δεδομένου ότι έχει τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της υπερασπών 10 του 2010. 330 εκατομμύρια για την ακρίβεια επέστρεψε η Κομισιόν στον τροποποιημένο προϋπολογισμό. Τώρα η Κομισιόν προτείνει να μην επιστρέψει αυτό το ποσό των 330. Αν δεν τα επιστρέψει τότε θα έχουμε περισσότερα ένα, ένα επιπλέον έσοδο το οποίο θα μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στον επόμενο προϋπολογισμό. Τι γίνεται τώρα με το πρόγραμμα ΙΤΕΑ με τη συμφωνία στην Κορεπέρ 1,3 εκατομμύρια χρηματοδότηση 750 εκατομμύρια προβλέπονται από, την, ε, από τον τίτλο 2, από την επικεφαλίδα 2. Είναι λοιπόν ένα περιθώριο το οποίο δεν υποχρεωθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το 2010 και σας εγγυώμαι ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε πια σήμερα γιατί το αγροτικό έτος έχει τελειώσει 15 Οκτωβρίου άλλα 269 εκατομμύρια προέρχονται από τη διάθεση περισσότερων πιστώσεων που μεταφέρονται το 2011. Τι θα γίνει τώρα, όταν θα έχουμε αυτά τα 330 θα ζητήσουμε λιγότερες, λιγότερη πίστοση. Λιγότερη πίστοση για τα προκυπευτικά και τις ενιαίες πληρωμές. Άρα λοιπόν το περιθώριο θα αυξηθεί το 2011 και έτσι θα έχουμε περιθώριο να χρηματοδοτήσουμε το ΙΤΕΑ. Αλλά αυτά τα 330 εκατομμύρια που κυκλοφορούν στο σύστημα, από αυτά τουλάχιστον 269 θα χρησιμοποιηθούν για το ΙΤΕΑ. Τώρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν δεν είχε εξαντλήσει τις πιστώσεις το 2010. Σωστό είναι ότι ξοδέψαμε λιγότερα. Αλλά θα αποζημιώσουμε για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου κράτη-μέλη 35% περισσότερα από πέρσι. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ξοδέψουν 35% περισσότερο το 2010 από ότι το 2009 για την ανάπτυξη της υπαίθρου. το οποίο μας ανησυχεί. Γιατί, διότι ε, δεν έχουμε ζητήσει όλο το ύψος του ποσού για το 2011. Πάντως συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις γι' αυτό και θα επανέλθουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή Λόγκο και να σας πω ότι Ανησυχώντας βέβαια για όλα αυτά, αλλάζουμε όμως θέμα και θα κλείσουμε τη σημερινή μέρα με δύο σημεία, το 5 και το 6 που θα τα συνεξετάσουμε. Είναι η τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεση στήριξη για τους γεωργούς, επιτροπολογία και εφαρμογή των ρυθμίσεων προσαρμογής στη Λισαβόνα θα ήθελα την κυρία Μογγέλ να τον κύριο Μογγέλ, συγγνώμη, να καλωσορίσω, διευθυντή τη Γενικής Διεύθυνση Γεωργία, που θα μα πει τι λεπτομέρειε για τη λογική της επιτροπή για την ευθυγράμμιση της νομοθεσία για τι άμεσε πληρωμέ και για θέματα ανάπτυξη της υπαίθρου. Ξέρετε ότι έχουμε μια σειρά 48 νομοθετικών προτάσεων προβλέπονται τις μήνες που ακολουθούν για να συμπληρώσουν αυτή την ευθυγράμμιση της γεωργικής νομοθεσίας το προσαρμόζοντάς το στην Λισαβόνα και τα θέματα αυτά για τη γεωργία είναι πολύ σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποφασίζεται η επιρροή και της δικής μας Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής και αυτό για τις πράξεις εφαρμογής της γεωργικής νομοθεσίας και το Κοινοβούλιο δεν επηρεάζει που δεν είναι τα πράγματα προς το παρόν. Στο γεωργικό τομέα ένα μεγάλο μέρος της εφαρμογής γίνεται μέσω της διαδικασίας διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 του 91 468 99-468 Συμβουλίου θα πρέπει να εξεταστεί όλο αυτό για να κάνουμε μια ταξινόμηση όλων αυτών των εφαρμοστικών πράξεων σύμφωνα με όσα ισχύουν μέσω της συνθήκης Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά να αποφασίσουμε αν πρόκειται για μια παραχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης είτε πράξεις εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 291. Να επιθυμίσω κάτι ότι για τις εξωμένες εκείνες πράξεις στο Κοινοβούλιο έχει δυνατότητα ελέγχου ιδιαίτερο, όπως ακριβώς και του Συμβουλίου, ενώ για τις πράξεις εφαρμόγης ε, δυστυχώς είναι πολύ περισσότερο περιορισμένε οι δυνατότητέ του. Αυτά ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικέ αυτά. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και τον Επίτροπο Σαντσόλους για το ε, ότι ξεκίνησε αμέσω αυτή την ε, εργασία ευθυγράμμιση. Ε, Μόγγελ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και ορισμένες διαφάνειες για να βοηθηθεί στην εισήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για το θέμα που έχετε ενώπιόν σας. Οι δύο πράξεις αφορούν την, το κανονισμό 73 του 2009 και το 698 του 2005 για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Λοιπόν, έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις Καταρχάς, στόχος μας είναι να ευθυγραμμίσουν την υπάρξη νομοθεσία βάσει των νέων απαιτήσεων της συνθήκης της Λισαβόνας για, τα, ε, για την, την εφαρμογή, την απαραίτητη εφαρμογή και δεύτερον να εισαγάγει στην νομοθεσία ε, τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία η Κομισιόν έχει αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν και νομοθετικό και συντακτικό θέμα. Όσον αφορά τώρα το θεσμικό ζήτημα, ε, θα παρουσιάσω καταρχάς τις επιπτώσεις στον, τομέα αυτό και εν συνεχεία θα με συμπληρώσουν συνάδελφοί μου για το θέμα της απλούστευσης. Τώρα, τι αλλάζει ουσιαστικά πριν από τη Λισαβόνα σε, βασικό, σε μια βασική νομοθετική πράξη η Κομισιόν είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει εφαρμοστικές πράξεις με λεπτομερούς κανόνες τους οποίους θα έχετε υπόψη σας από, από το παρελθόν. Και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου ήταν ότι η Κομισιόν ενεργούσε βάσει της διαδικασίας επιτροπολογίας χωρίς την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Στο πλαίσιο των βασικών νομοθετικών πράξεων η Κομισιόν έχει την δυνατότητα πρώτον να υιοθετήσει και εν συνεχεία να εξουσιοδοτήσει πράξεις Μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει και να εφαρμόσει πράξεις. Όσον αφορά λοιπόν την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των πράξεων, η συνθήκη της Λισαβόνας βάσει το άρθρο 291 δίνει την ε, εξουσία στην Κομισιό να υλοποιεί αυτές τις πράξεις. Όσον αφορά τώρα την ανάθεση, ανάθεση εξουσιών, τι λέει το άρθρο 290. Λέει βασικά ότι μια νομοθετική πράξη μπορεί να αναθέτει στην Κομισιό την ισχύ υιοθέτηση ε, μη νομοθετικών πράξεων ή γεν, γενικής εφαρμογής ή να συμπληρώνει ή τροποποιεί ορισμένε μη ουσιαστικέ πτυχέ νομοθετικών πράξεων. Το άρθρο λοιπόν 290 δίνει και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο νομοθετικών πράξεων και λέει ότι ουσιαστικά στοιχεία των νομοθετικών πράξεων διατηρούνται στα χέρια του νομοθέτη βάσει της ε, συνθήκης. Το άρθρο 290 επίσης καθορίζει ότι η έλεγχοι ε, τα δικαιώματα ελέγχου που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ορίζονται από τη συνθήκη και επίσης ε, η ανάθεση αυτών των πράξεων δεν μπορεί να τεθεί ενισχύ πριν περάσει η περίοδος ε, τυχόν αντιρρήσεων που, πρέπει να, που, που θα υποβληθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο αντιρρήσεων ε, και άμα περάσει αυτό τότε μπορούν να τεθούν ισχύ. Τώρα εφαρμοστική ισχύς. Άρθρο 291. Εκεί λέει ότι τα κράτη-μέλη θετήσουν όλα τα μέρη της εθνικής νομοθεσίας που χρειάζονται για να εφαρμοστούν ε, νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης. Το 2, η παράγραφος 2 λέει όπου υπάρχουν ενιαίες συνθήκες εφαρμογής, η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει εφαρμοστικές πράξεις και αυτό συμβαίνει, θα συμβεί όταν υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε ακριβώς αυτές τις ομοιόμορφες συνθήκες ε, εφαρμογής. Πρέπει λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε μία ομοιομορφία στην διαδικασία εφαρμογής των νομικά θεσμευτικών πράξεων. Τα δικαιώματα ελεγχού των κρατών μελών δεν ορίζονται στη συνθήκη, αλλά θα καθοριστούν σε ένα συγκεκριμένο κανονισμό, ο οποίος συζητείται τώρα, το ανέφερε και ο Πρόεδρος, και έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα νομοθεσία επιτροπολογίας. Και πάλι ε, αυτές οι εφαρμοστικές πράξεις ορίζονται στις λεπτομέρειες ε, του εφαρμοστικού τμήματος της πράξης. Ευθυγράμμιση. Τι εννοούμε με ευθυγράμμιση. Ο στόχος του άρθρου 290, ε, του 290 είναι να δώσει στον νομοθέτη όλες τις δυνατότητες που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας για την ανάθεση ε, πράξεων. Ε, σας είπα ότι οι δύο αυτοί κανονισμοί, έχουμε δύο προτάσεις για ευθυγράμμιση, είναι ο κανονισμός 73-209 άμεσες πληρωμές και 1698 του 2005 για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Για την ευθυγράμμιση ληφτών θα ακολουθήσει μια σειρά κειμένων με τις προτάσεις και για, την, για τις δημοσιονομικές πτυχές και για τη διαμόρφωση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Περίπου 50 προτάσεις πρέπει να γίνουν, μπορεί λίγο να μειωθεί ο ρυθμός αυτός, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι λιγότερες πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή με τη νέα συνθήκη. Ποιε είναι οι βασικές αρχές όλη αυτής της άσκησης, ευθυγράμμιση, Καταρχάς είναι να υιοθετήσουμε το κεκτημένο, να, να προσαρμόσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στη συνθήκη της Λισαβόνας. Λοιπόν, να προσαρμοστούμε στη συνθήκη. Ε, η συνθήκη αυτή δεν δίνει, και το τονίζω, δεν δίνει πρόσθετες εξουσίες στην Κομισιόν. Ο στόχος λοιπόν της ευθυγράμμισης είναι να ε, μοιράσουμε τις υπάρχουσες εξουσίες της Κομισιόν σε δύο σκέλη Καταρχάς, επί της βάση ενός μελετημένου screening των βασικών πράξεων, μιας πολύ εμπεριστατωμένης δηλαδή εξέτασης των βασικών ε, πράξεων, για να μπορέσουμε να επισημάνουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εδρεωθεί μέχρι τώρα και εν πρέπει να μελετήσουμε όλα το, το υπάρχον και εκτιμένο για να μην χαθούν πράξεις οι οποίες είναι μίζωνος σημασίας. Και δεύτερον, να καθορίσουμε αντικειμενικά νομικά κριτήρια για την εφαρμογή των νέων πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι οι στις εξουσίες της Κομισιόν πρέπει να μοιραστούν καταρχάς στις κατεξουσιοδότηση εξουσίες και στις εφαρμοστικές εξουσίες, όπως αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια για, αυτή την, ε, για αυτές τις εξουσίες, τις κατεξουσιοδότηση και τις εφαρμοστικές. Άμα δείτε το κείμενο του άρθρου 290, όταν λέμε delegated, κατεξουσιοδοτηση πράξη πράξης μη νομοθετικέ, δηλαδή έχουν γενική εφαρμογή, μοιάζουν με νομοθετήματα ε, και ε, τροποποιούν ή συμπληρώνουν νομοθετικέ πράξεις. Ε, εν συνεχεία, το άλλο σκέλος, εφαρμοστικές, εκτελεστικές εξουσίες, σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση, για την εφαρμογή και ότι το άρθρο 290 έχει ως στόχο την ουσία των νομοθετικών αποφάσεων, ενώ το 291 στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή αυτών των πράξεων. Πώς τώρα θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες πράξεων. Καταρχάς υπάρχουν δύο ε, παραδείγματα που μπορούμε να κάνουμε μία, ένα σαφή διαχωρισμό. Καταρχάς, σα, σαφής ε, κατανάσταση, κατεξουσιοδότηση εξουσίας είναι πράξεις γενικής εφαρμογής που έχουν ως στόχο την τροποποίηση νομοθετικών πράξεων. Ε, όταν γίνεται προσπάθεια ευθυγράμμισης, αυτές οι πράξεις πρέπει να οριστούν ως delegated acts, δεδομένου ότι ο στόχος τους είναι να τροποποιήσουν οι υπάρχουσες νομοθετικές πράξεις. Όταν λέμε τώρα καθαρά για εφαρμοστικές εξουσίες, εννοούμε πράξεις με μονομένης ε, εφαρμογής, οι οποίες ε, χρειάζονται για την ενιαία εφαρμογή από τα κράτη-μέλη της πράξης αυτής. Δηλαδή, με μονομένες εφαρμογές για την υιοθέτηση μιας πράξης από ένα κράτος μέλος. Υπάρχει λοιπόν μια οριοθετική γραμμή για άλλες πράξεις γενικής εφαρμογής είτε ε, όταν συμπληρώνουν τις νομοθετικές πράξεις ή όταν χρειάζονται για μία ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε, να υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να ξεχωρίσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες. Πρώτον πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε το κέντρο βαρύτητας των μέτρων. Δηλαδή εάν ένα μέτρο αναφέρεται στο περιεχόμενο, μια πράξη αναφέρεται στο περιεχόμενο μιας ε, νομοθετικής απόφασης, τότε ο νομοθέτης ε, έχει στα χέρια του μία κατεξουσιοδότηση πράξη. Όταν όμως ε, το περιεχόμενο έχει σχέση με εφαρμοστικά μέτρα, τότε μιλάμε για εφαρμοστική πράξη. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα πριν μπω στις λεπτομέρειες. Όταν λέμε κάτι εξουσιοδότηση πράξης, εννοούμε πράξεις ε, όπου συμπληρωματικές ε, προδιαγραφές καταλληλότητος ορίζονται ε, όταν στήθενται ορισμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει οι γεωργοί παραδείγματος χάρη να τηρούν για να λαμβάνουν ενισχύσεις ή όπου συμπληρώνουμε ορισμούς στο παρελθόν π.χ είχαμε διαφορετικούς ορισμούς για τις ε, αρρώσιμες εκτάσεις, παραδείγματος χάρη. Άλλος ήταν ορισμός στο Συμβούλιο, άλλος ήταν ορισμός στην Κομισιό. Ε, επίσης, ε, ο ορισμός υποχρεώσεων ελέγχου, ο ορισμός των κυρώσεων και οι απαιτήσει εγγύσεων είναι μια, ένα κριτήριο που είναι αναγκαίο, μια προδογραφή αναγκαία για την εσωτερική αγορά. Οι προτάσει ευθυγράμμιση για τι άμεσε πληρωμέ στον κανονισμό 73-2009 θα καλύψουν τρει τρεις ε, διατάξεις κάτω εξουσιοδότηση πράξεων, τις οποίες βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Άρθρο 45α1, που αναφέρεται στις, ε, ε, στους κανόνες επιλεξιμότητος και όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν οι προδιαγραφές και τα κριτήρια. Διότι πλέον εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα. Ε, το άρθρο 45α3 που αναφέρεται στα, στις, στα κληροδοτήματα, στις κληρονομιές όταν κληρονομείται μία εκμετάλλευση και όπου υπάρχει τίθεται θέμα άμεσων πληρωμών. Και τρίτον, ε, στις κατεξουσιοδότης πράξης είναι το άρθρο 45α5 που αναφέρεται στην καταβολή άμεσων πληρωμών όταν χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι σπόροι ε, για πιστοποιημένες καλλιέργειες. Και αυτό ανήκει λοιπόν στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Και ορισμένα παραδείγματα των εφαρμοστικών πράξεων. Εδώ αναφέρομαι στις λεπτομέρειες της διαδικασίας εφαρμογής. Παραδείγματο χάρη, ποια έγγραφα, ποια έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν, ποιες ε, ρυθμίσεις ελέγχου εφαρμόζονται, πρακτικές ρυθμίσεις για έγκριση προγραμμάτων, πληροφόρηση, υποχρέωση πληροφόρησης, τι πληροφορίες ε, πρέπει να δώσουν στις εθνικές αρχές και εν συνεχεία στην Κομισιόν και τέλος ε, εκθέσεις, αναφορές. Υπάρχουν υποχρεώσεις ε, υποβολής εκθέσεων, αναφορών σε αυτό το πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό 73 έχω γράψει, είναι λάθος η διαφάνεια, αναφέρομαι στον κανονισμό 73 και άρθρο 27β. Άφορα α, τις ποιοτικές προδιαγραφές για να καταγραφεί η ταυτότητα του παραγωγού. Το άρθρο 33.6 αναφέρεται στην, στην εφαρμογή των δικαιωμάτων, του πλαισίου δικαιωμάτων, όταν τα δικαιώματα του παραγωγού δεν έχουν ακόμα απολύτως καθοριστεί. Και το 41.7 φορά τα δικαιώματα καταβολής πληρωμών, όταν ο παραγωγός δικαιούται να λάβει ορισμένες πληρωμές σε βάση δικαστικής απόφασης. όλα αυτά είναι εφαρμοστικές πράξεις. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, πιστεύω ότι το κέντρο βάρους, όπου το κέντρο βάρους είναι στην ομοθετική πλευρά, θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Όπου το κέντρο βάρους βρίσκεται στο διοικητικό, στη διοικητική πτυχή των κρατών μελών, εκεί οι πράξεις θα έχουν τη φύση εφαρμοστικών, τη μορφή εφαρμοστικών πράξεων. Και τώρα θα σας αναφέρω ορισμένα άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά ολοκληρώνοντας. Όπως είδατε στην αρχή, πρέπει τα κείμενα να καθορίζουν τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της ε, παραχώρησης, του delegation. Ε, ε, ε, και αυτά καθορίζονται ακριβώς. Όμως στις δύο αυτές προτάσεις δεν είπαμε τίποτα για την διάρκεια αυτών των κατεξουδότησης πράξεων. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί και στις δύο περιπτώσεις και στην ανάπτυξη πέθρου και την απευθείας πληρωμές αναγκαστικά υπάρχει περιορισμός με την προγραμματική περίοδο πενταετίας, δηλαδή το 2013. Άρα δεν έχει νόημα τώρα να πούμε ότι η διάρκεια ζωής θα είναι πενταετής αν γνωρίζουμε ότι προηγουμένως ε, ήδη θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Έτσι και αλλιώς. Δεύτερο σημείο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, πρέπει να έχουν έλεγχο του μέτρου της Κομισιόν μετά την έγκρισή του. Και δύο είναι τα πιθανά μέσα. Η ανάκληση της ε, εξουσιοδότησης ή αντίθεση. Ανάκληση της εξουσιοδότησης σημαίνει ότι κάθε κλάδος του, του νομοθετικής εξουσίας, κοινοβούλιο ή ε, συμβούλιο, μπορεί να άρει αυτή την εξουσιοδότηση από την Κομισιόν. Αυτό δεν βλάπτει την πράξη που έχει εγκριθεί, αλλά δεν μπορεί πλέον η Κομισιόν να εγκρίνει περαιτέρω πράξεις. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει το δικαίωμα της νομοθετικής αντίθεσης που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να αντιταχθούν σε μια πράξη τη Κομισιόν που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί αυτή να τεθεί εν ισχύ. Δηλαδή και οι δύο δυνατότητε ελέγχου έχουν ενσωματωθεί στι δύο αυτέ προτάσει. Θα διαπιστώσετε δηλαδή ότι και το δικαίωμα αντίθεση και το δικαίωμα ανάκληση περιλαμβάνεται στα κείμενα αυτά. Το τελευταίο σημείο που θέλω να θέσω είναι ότι φυσικά δεν υπάρχει πλέον στο πλαίσιο των κατεξουδότηση πράξεων ψηφοφορία ε, από την Επιτροπή. Δεν προβλε... από επιτροπή. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ε, ε, ε, δηλαδή η Κομισιόν εγκρίνει χωρίς οποιαδήποτε επιτροπολογία. Θα υπάρξει όμως η οργάνωση από την Κομισιόν μια ολόκληρης διαδικασία προετοιμασία που θα συνεπάγεται αφενός με ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου την διαβούλευση με εμπειρογνώμονες που εν γέννη θα προέρχονται από ε, τα κράτη-μέλη, αλλά βεβαίως πρόσβαση θα έχει εκεί και το ε, Κοινοβούλιο. Θέλω επίσης να επισημάνω το, τη Συμφωνία Πλαίσιο που μόλις ενέκρινε η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν δύο μέρες. Στο ε, άρθρο 15 προβλέπεται ότι η Κομισιόν θα παράσχει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συναντήσεις με εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της δουλειάς της για την εφαρμογή και προετοιμασία νομοθεσίας της Ένωσης και του ίδιου δικαίου και των καταχώρηση πράξεων ε, και μπορεί να, να παρακαλέσει ε, να καλέσει και εμπειρογνώμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει. Έτσι δείχνει με ποιο τρόπο μπορεί ή θα μπορούσε να εμπλακεί το Κοινοβούλιο στην όλη αυτή διαδικασία τη προετοιμασία. Αυτά θέλω να σα τα πω για, στα πλαίσια τη γενική ενημέρωση ε, σχετικά με τη διαδικασία ευθυγράμμιση, κυρίω σε σχέση με του δύο κανονισμού που έχουν προταθεί για τι άμεσε πληρωμέ και την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα θα ζητήσω από τους ε, συναδέλφους να σας ε, παρουσιάσουν τα ουσιαστικά σκέλη αυτής της πρότασης που αφορούν την εφαρμογή. Παρακαλώ σύντομα σύντομα όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα παρουσιάσω εν συντομία δύο μικρές αλλαγές ε, στον κανονισμό, που, αλλαγές που είναι ουσιαστικές. Την πρώτη, η πρώτη αφορά το άρθρο 19.1, το σημείο 9 της πρότασης. Ε, ε, προστίθεται μια νέα υποπαράγραφος, ένα νέο εδάφιο. Η πρώτη, ε, το πρώτο εδάφιο αφορά την, την ευθυγράμμιση και έχει μετα... είναι η μεταφορά των εφαρμοστικών κανόνων. Αλλά η δεύτερη... το δεύτερο εδάφιο ε, αφορά την πρόταση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο πέρσι. Και υπάρχει και μια απλούστευση, πρόταση απλούστευσης που προκύπτει από τις 39 αυτές προτάσεις και αφορά την ε, δήλωση της ε, έκτασης. Εν γέννη, όλοι οι ε, οι καλλιεργητές, όλοι οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν όλες, όλα τις, ε, τα εδάφη τους και πρέπει να το επισημάνουν σε ένα χάρτη που πηγαίνει στις εθνικές αρχές. Θέλουμε να πούμε ότι ε, για ε, τους παραγωγούς που δεν ζητούν ενίσχυση που να ε, εξαρτάται από τις εκτάσεις και αν οι εκτάσεις που κατέχουν δεν ξεπερνούν το ένα εκτάριο δεν χρειάζεται να κάνουν τη δήλωση. Πρέπει όμως να υποχρεωτικά να δηλώσουν εάν έχουν τέτοια αγροτική γη και αυτό οφείλεται στην πολλαπλή συμμόρφωση και ε, στις ε, περιβαλλοντικές συνθήκες, συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος. Γι' αυτό πρέπει οι αρμόδιες αρχές να γνωρίζουν εάν έχουν αγροτικές γης η παραγωγή αυτή ή όχι. Τέλος υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο άρθρο 21.1 που δεν έχει άμεση σχέση με την απλούστευση. Είναι μια παράληψη που έγινε κατά τον έλεγχο υγείας. Το άρθρο 28 αφορά τις ε, μήνυμες απαιτήσει για την καταβολή της άμεσης ενίσχυσης. Αυτό μπήκε κατά τον έλεγχο υγείας, το health check. Τώρα η Κομισιόν μπορεί είτε να θέσει ένα ε, όριο εκταρίων ή ένα όριο ποσού το 28.1 ε, έχουμε, αφορά την περίπτωση που το κράτος μέλος έχει επιλέξει το ε, κατόφλιο εκταρίων, ε, της, των εκτάσεων και ε, προβλέπει ότι πρέπει μπορούν να ε, ξερούνται οι ε, μικροί, μικροί γεωκτήμονες. Ακόμα και ο κανονισμός 73 ή οι εφαρμοστικοί κανόνες του 1120 του 2009 αποδέχονται την αναφορά στη συγκεκριμένη ενίσχυση, το λεγόμενο μέτρα άρθρο 68. Αυτά έλειπαν πριν και τώρα προστέθηκαν στο άρθρο 28, παράγραφος 1. Αυτές είναι όλες οι τροπολογίες που αφορούν την άμεση ενίσχυση. ευχαριστώ. Θα συνεχίσω σύντομα όσον αφορά την απλοποίηση αυτού του ενδεχόμενου του όρου ε, στην πρόταση αυτή και σύμφωνα με τα 23 και 24 άνθρωπα που προτείνονται και μετά από τις 39 προτάσεις μιας ομάδας κρατών μελών και για τον υποθετικό αυτό χαρακτήρα, τον δυνάμει, τον δυνάμει χαρακτήρα, θα δούμε τις δυνατότητες να αλλάξουμε τον κανονισμό 73 του 2009. Εδώ πρόκειται για την απλοποίηση αυτής της παρακολούθησης ε, σε περιπτώσεις που δεν συμφωνούν ε, σύμφωνα με τον κανόνα του ελαχίστου ή το, ε, την ελάχιστη μη συμμόρφωση και όπως έχει σημαίνει τα πράγματα. Εάν δεν υπάρξει κάτι που να συμφωνεί με αυτό με μια μείωση ανακτέρω των 100 ευρώ είτε τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι λόγω του εύρους αυτού του φαινομένου που αυτή η μη συμμόρφωση είναι ελάχιστη, τότε σύμφωνα με τη σημερινή ρύθμιση τα κράτη-μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν άμεσα μια μείωση της ενίσχυσης στο Γεωργό, αλλά να δώσει στο Γεωργό τη δυνατότητα να την προσφέρει σε μια κάποια προθεσμία, σε μια ε, βοήθεια, ε, ε, μια ενίσχυση, μια ενίσχυση η μη συμμόρφωση και αυτό υπέρ του Γεωργού λοιπόν εγώ σας περιέγραψα τη σημερινή ρυθμίση είναι υπέρ του Γεωργού αλλά με κάτι το αρνητικό όμως οι υπηρεσίες ελέγχου κατά τρόπο κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένε να ασκούν ένα έλεγχο σε όλους τους Γεωργούς οι οποίοι, για τους οποίους ακριβώς εφαρμόστηκε αυτός ο κανόνας του ελαχίστου. Και αυτή η απλοποίηση όπως προτείνουμε στο κείμενο μας επιτρέπει έτσι αυτή η έλεγχη που να διαπιστώνουν αν έχει αλλάξει τα πράγματα ο Γεωργός ή όχι, όλα αυτά να γίνονται όχι κατά σημαντικό τρόπο ετησίως σε όλους αυτούς τους Γεωργούς, αλλά να μπορεί να προχωράει κανείς σε μια δειγματοληψία, δηλαδή τα κάτι μέλη να δουν μια ανάλυση του κινδύνου και να ασκήσουν αυτόν τον έλεγχο, αυτές τις... Ε, ε, τις ε, επισκέψεις σε εκείνους που παρουσιάζουν αυτή τη δυνατότητα ότι ίσως δεν διόρθωσαν τα πράγματα. Εντάξει, προς το παρόν από το σημερινό κείμενο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Και μια ελάχιστη μεταβολή του εγγράφου, θα το πω στα αγγλικά που είναι το πρωτότυπο κείμενο, το ensure από το verify αντικαθιστώ με το με, και της απονομικής πλευράς ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια παρόμοια ε, εξουσιοδότηση, ας το πούμε έτσι, για αυτή τη δυνατότητα ελέγχου μέσω ορισμένων μονομένων περιπτώσεων δειγμάτων. Αυτό λοιπόν σχετικά με αυτή την πολλαπλή συμμόρφωση και ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν επιτρέπετε, ο κύριος Πίλκε θα ολοκληρώσει με την ειδική πρόταση που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Υπέθρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την ανάπτυξη υπαίθρου, ε, σκεφτόμαστε να υποβάλουμε τις εξής προτάσεις. Πρώτον, θα μειώσουμε τον αριθμό των ε, ε, εκθέσεων στρατηγικής, ανακεφαλικών εκθέσεων στρατηγικής που πρέπει να υποβάλουν τα κράτη-μέλη από 3 σε 2 το 2013 και το 2015. Δεύτερον, η, παρακολούθηση της ομάδας υψηλού επίπεδου για το γάλα μάλλον σε συνέχεια της εργασίας της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για το γάλα και ε, υπό το φως της διατροφικής αλυσίδας ε, και τα 27 κράτη-μέλη θα έχουν τέτοιες ομάδες. Δηλαδή το μέτρο θα διατίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη πέθρου και θα και θα μπορούν να ενισχύονται οι ομάδες παραγωγών ε, ε, στο πλαίσιο του καθεστώτος οργάνωσης αγοράς ε, απορροκυπευτικών. Ενώ τώρα αυτό δεν είναι δυνατόν. Επιπλέον, θα φτιάξουμε μία κατά περίπτωση εφαρμογή του μέτρου της χρήσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον παραγωγό. Ε, υπάρχει μια ελάχιστη υποχρέωση δηλαδή. Πρέπει ο παραγωγός να ενημερωθεί για την πολλαπλή συμμόρφωση. Οι συμβουλές μπορεί να ε, συμπληρώνονται από άλλες που είναι σημαντικές γιατί συγκεκριμένη ε, μονάδα. Τώρα, όσον αφορά τις, τις πληρωμές για την περιοχή Natura 2000, είναι επιλέξιμες οι περιοχές που συνδέουν περιοχές Natura 2000 και που είναι σημαντικές για περιβαλλοντικά ωφέλη ε, και εισφέρουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας για τους βιοτόπους γιατί το βασικό μας, ο βασικός μας σκοπός είναι οι καθορισμένες περιοχές Natura 2000 αλλά και αυτές οι περιοχές έχουν περιβαλλοντική αξία και γι' αυτό θα εξασφαλίσουμε την ε, περιορισμένη επιλεξιμότητά τους. Επιπλέον, θα κάνουμε μία μελέτη επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση κάποιων περιοχών, δηλαδή θα εισάγουμε ε, το στοιχείο του κινήτρου που ήδη περιλαμβάνεται σε άλλα σημεία της νομοθεσίας. Δηλαδή το κόστος θα είναι επιλέξιμο μόνον όταν έχει γίνει αίτηση για το μέτρο. Η επιλεξιμότητα λοιπόν ξεκινά μόνο όταν έχει δοθεί η αίτηση. Όσον αφορά τις, ε, ε, ε, τις παραβιάσεις μίζωνος σημασίας, δίνω το λόγο στον άδελφο. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε τώρα να διευκρινίσουμε όλο αυτό το σύνολο πληροφοριών που μας προσέφεραν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Ε, τον ε, Διευθυντή Μέγκελ θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί με σαφήνιζε μας παρουσίασε αυτό το θέμα με το οποίο ασχολούμεθα την ευθυγράμμιση με την συνήθεια της Λαβώνας της ρύθμισης της γεωργικής και τη δυνατότητα σε κάθε περίπτωση μεμονωμένα να αποφασίσουμε για την εφαρμογή του άρθρου 290 πράξεις εκτελεστικές και 91 τις κατεξιδότηση πράξη. και να καθορίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου επίσης και στις εφαρμοστικές πράξεις και ίσως βέβαια ναι, και τις δυνατότητες μεταβολής των πράξεων αυτών των νομοθετικών σύμφωνα και με τη Λισαβόνα για να προβούμε σε απλουστεύσει, απλοποιήσεις όπως το είπαμε να μπορεί κανεί να παρέμβει στην όλη ρύθμιση για να διορθώσει και να απλοποιήσει εκεί που είναι δυνατό. Ε, σημαντικότατο βέβαια είναι στην, ε, όπως μας είπε πολύ καλά ο ε, διευθυντής στην ε, διαχωρισμό ανάμεσα στην ε, κατοξιοδότηση και των υπολείπων να καθοριστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου που σύμφωνα και με τη Σταβόνα δεν είναι μόνο μια πρωτογενής νομοθεσία έτσι τη στιγμή ακριβώς που πλάθουμε τον νόμο αλλά